Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να αρχίσουμε τη συνεδρία. Συζητώ συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Και όπως είχαμε συμφωνήσει εχθές στην έναρξη των εργασιών μας, σας προτείνω να ασχοληθούμε αμέσως με το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση κυρίας Κορνέλησεν Συγκεκριμένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών για το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας. Το λόγο έχει η συγκεκριά, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Έχω εργαστεί εκτατικά και εντατικά τα τελευταία χρόνια, δύο χρόνια για τα Βαλκάνια και είδα τι μπορούν να κάνουν τα προενταξιακά κονδύλια και τι δεν μπορούν βεβαίως να κάνουν. Για να προσανατολιστώ, συζήτησα με πολλές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικούς εταίρους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, άλλους ενεχομένους και με την εμπειρία αυτή και την ενημέρωση που απεκόμισα έκανα κάποιες αλλαγές στο κείμενο ένα σημαντικό σημείο ήδη είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, υποψήφιες χώρες και προϋποψήφιες για την επιλεξιμότητα από το μέσο προενταξιακής βοήθειας. Τώρα αλλάζει αυτό για τη βοήθεια για την απασχόληση και κοινωνική πρόνοια είναι ήδη επιλέξιμες με τον τρόπο αυτό. Τι άλλαξα λοιπόν στο εγγραφό μου. Νομίζω ότι τα χρήματα του προεταξιακού μέσου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την ενίσχυση των επενδύσεων και διεθνώς αλλά και ε, χωρίως και οι φραγμοί που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών θα πρέπει να καταργηθούν. Τι εννοώ capacity building, ε, περιφερική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική απασχόληση, εδαφική ε, συνεργασία και περιφερειακή. Προς το παρόν, τα περισσότερα χρήματα ε, είναι σε ξεχωριστές συνιστώσεις και δεν μπορούν να συνδυάζονται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε χάνουν ευκαιρίες οι χώρες αυτές. Παράδειγμα, θα ήθελα ας πούμε ένα εργοστάσιο να φτιαχτεί ένας δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο μέχρι την επιχείρηση. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν χρήματα από το προενταξιακό μέσο για να απασχολήσουν τον τοπικό πληθυσμό και να τον εκπαιδεύσουν, να τον καταρτήσουν, να φτιάξει το δρόμο. Επίσης, ε, συμπεριλαμβάνω και το θέμα του φύλου και των ε, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όχι μόνο στην κοινωνική διάσταση αλλά και αλλού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, για τη γεωργία και την ανάπτυξη της Ενίσχυσε επίσης το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και την ανάγκη ακριβώς να δημιουργούνται οι δυνατότητες για ε, εργοδοτικές οργανώσεις και συνδικάτα για να μπορούν να συμμετέχουν τελικά και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο. Διότι αυτή τη στιγμή σε πολλές υποψήφιες χώρες Τα συνδικάτα γνωρίζουν ε, τουλάχιστον την καχυποψία του κόσμου, ενώ οι εργοδοτικές οργανώσεις συχνά ε, δημιουργούν καρτέλ κοινωνικοί εταίροι στο πρωταξιακό μέσο δεν έχουν ειδική μεταχείριση. Θεωρούνται άλλη μια κοινωνική οργάνωση, κοινωνική ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστή προσοχή. Η κοινωνία των πολιτών είναι βεβαίως ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο για να δημιουργηθεί πραγματική δημοκρατία. Αυτό το τόνισα στην ε, γνωμοδοτησή μου. Και επίσης και το δικό μας ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Um, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτήσει προσεχώς ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το προενταξιακό μέσο και ε, να το κάνει πιο συνεκτικό και πιο αποτελεσματικό και θα πρέπει να το καλωσορίσουμε κι εμείς, αλλά και η κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπόνηση καν αυτού του εγγράφου. Είπα επίσης ότι εκθέσεις προόδου για τις χώρες στις οποίες ε, αφιερώνουμε πολύ χρόνο, πολύ κόπο και πολύ προσοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη θα ψηφίσουμε μερικές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των ε, γράφων στρατηγικής για τις ε, εκάστοτε χώρες. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να τονίσω ως αλλαγή. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι οι χώρες σιγά σιγά θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση ε, της βοήθειας μόνες τους καθώς δημιουργούν τις υποδομές. Και πρόσθεσα να συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή αν οι πολιτικές αποφάσεις σε μια χώρα ή ο τρόπος που λειτουργεί η διοικητική μηχανή της φθήνουν, ας πούμε, λόγω πολιτικών διαπλεκτισμών, μποϊκοτάζ του Κοινοβουλίου ή άλλων προβλημάτων, θα μπορούσε ενδεχομένως να τους αφαιρείται και η διαχείριση. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία μας με τους κοιοδησηγητές και να ακούσω τώρα τις προτάσεις σας και τις ε, απόψεις. κυρία Στάιρουκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, είναι πάρα πολύ καλή η έκθεσή της γνωμοδότηση μάλλον, και πολύ νωρί συμπεριέλαβε και τι δικέ μα προτάσει. είναι σημαντικό ότι τονίζει και ενισχύει και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις και βαθιές αλλαγές στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη. Καλωσορίζω την πρόταση που κάνει η συγγήτρια. 1,5% της οικονομικής βοήθειας να πηγαίνει στους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορώ παρά να το υποστηρίξω αυτό εξ ονόματος της ομάδας μου. Άλλο θέμα. Η προενταξιακή βοήθεια θα πρέπει να δίνεται στις χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουν ερωτηθεί οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν ακριβώς γιατί αυτή η ομάδα δεν είχε συμπεριληφθεί αρκετά στην εκπόνηση των προγραμμάτων. Ενίσχυση λοιπόν των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου. Επαφή λοιπόν μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των ε, κοινωνικών εταίρων είναι κάτι το οποίο μπορεί να προωθηθεί και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις του χώρου. Και όταν δημιουργούνται νέα κοινωτικά προγράμματα θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη ενημέρωση με ειδικέ εκδηλώσεις για τις ομάδες αυτές, γιατί πολύ συχνά η αποτυχία δεν οφείλεται στην έλλειψη ενθουσιασμού, η δέσμευσης η στράτευση του πληθυσμού, αλλά σε έλλειψη προφόρησης λόγω κρατικών αδυναμιών και προβλημάτων οργάνωσης. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ την συγκήτρια και χαίρομαι για την έκθεση της, οποία και καλώς Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Αυτή ήταν η συζήτηση. Ροζ κόκκινη. Όχι, τι λέω ροζ κόκκινη. Πράσινη και κόκκινη. Η πράσινη. Εν πάση περιπτώσει με τη σειρά που θέλετε. Η συγγήτρια, παρακαλώ. Well, yes, I'd to. Μάλιστα. Τι θέλετε να ολοκληρώσω, να μακρηγορήσω για να έρθουν και άλλοι να μιλήσουν. Ευχαριστώ την κυρία Στάιμπλ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πλήρη της υποστήριξη. Πιστεύω αυτό το θέμα της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικότατο. Καταναλώσαμε πολύ κόπο και πολύ χρήμα για να οικοδομήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι αναγκαίες διαδικασίες από τις κρατικέ αρχέ για να συμμετέχουν οι ενεχόμενοι. Λοιπόν, τι νόημα έχει να έχει στηθεί μια κοινωνία των πολιτών. Αναφέρθηκε στο 1,5% τη χρηματοδότηση. Να σταθώ λίγο εδώ. Εδώ και χρόνια ήταν πάγια υπόσχεση ότι τα χρήματα που αφιερώνονται στην κοινωνία των πολιτών θα διπλασιαζόντουσαν. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα το ποσό. Αφιερώσαμε εμείς και χρόνο στον υπολογισμό του ποσοστού που θα πρέπει να είναι τώρα, γιατί συνολικά τα κονδύλια αυξάνονται. Δηλαδή, αν διπλασιάζαμε τα κονδύλια της κοινωνίας των πολιτών θα έβγαινε τελικά 1,5%. Αυτό θα συζητηθεί και τελικά θα διευθετηθεί στην ίδια την Επιτροπή Εξωτερικών που είναι καθήλια αρμόδια, αλλά θα πρέπει να στείλουμε αυτό το ισχυρό μήνυμα. Εγώ προσβλέπω συνεργασία μου παρόλα αυτά και με τους υπόλοιπους όδης Ευχαριστώ. 2 Απριλίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για, την, ε, για τις τροπολογίες. 23 και 24 Απριλίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Στις 31 Μαΐου ε, θα τις εγκρίνουμε και θα αφήσουμε την ΑΦΕΤ στις 7 Ιουνίου να αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη τη δική μας γνωμοδότηση. Ολοκληρώσαμε για αυτό το σημείο ναι. και διακόπτω τώρα μέχρι τις 9.30 που θα έρθουν οι συνάδελφοι για να ψηφίσουμε. Ζητώ συγγνώμη όλος ιδιαίτερος τους διερμηνείς. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer parce que les rangs se sont remplis. Αγαπητοί συνάδελφοι, μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Βλέπω ήρθατε όλοι, οπότε δεν χρειάζεται να καθυστερούμε άλλο. Όπως σας είπα χτες στην αρχή των εργασιών μας, θα αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Α, ωραία ησυχία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ε, ψηφοφορία για το σημείο 13, δηλαδή την γνωμοδότηση της κυρίας Τσίμερ για την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, της Επιτροπής ε, των Γυναικών για την εφαρμογή της αρχής της, ισότητας, της μισθολογικής ισότητας για άνδρες και γυναίκες για την ίδια εργασία. Παράγραφος 1, συμβιβαστική α ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 5. Η συγκήτρια προτείνει αποχή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές. Δεν ψηφίσατε όλα, αλλά έχω την εντύπωση πως εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβαστική β, τέσσερα, τεσσάρων ομάδων με μια προφορική τροπολογία που υποβλήθηκε γραπτός. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε για την ε, Β λοιπόν. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική για την ε, συμβαστική Β. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Tout le sa carte Non, non, alors dites-moi, dites-moi, dites-moi, qui n'a pas sa carte Ποιος δεν έχει κάρτα, για να μου πει. Λοιπόν, δεν έχω κλείσει ακόμα την ψηφοφορία. Μπορείτε να βάλετε την κάρτα σας τώρα. Tout le monde Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 24 κατά. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα επαληθεύσουμε, ναι, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν ε, φάνηκε καλά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 32 κατά. Απορρίπτεται. Et quoi, quoi, attendez. Euh, bon, allez, l'amendement 7 de Madame Hirsch. Qui est... 7 της κυρίας Hirsch τώρα με τις 8 και 9 που είναι ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ των τριών αυτών τροπολογιών. Κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 7, 8 και 9. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 22 κατά, λέει η πρόεδρος. Αν είναι το αντίθετο είναι 22 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καταπίπτουν. Όχι, η 11 είναι συμβατή. Μάλλον όχι, όλες είναι συμβατές. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 του κυρίου Μπεναμιάς ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 Νταρντέν υπέρ Δώδεκα καταπίπτει. Και ψηφίζουμε μετά την παράγραφο 2 την τροπολογία 13 της κυρίας Πλάμ. Η συγκίτρια είναι απέχει, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 Μάκιντάερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 τις εισηγήτριες υπέρ 17 υπέρ ποιοι είναι 17 ποιοι είναι υπέρ Ναι, αλλά δεν ε, ψήφισαν μαζί σας ε, οι ΕΣΕΡ. Εγώ εντάξει, ναι, να ελέγξω όταν υπάρχει αμφιβολία. 17, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική γάμα σε από 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 24 της κυρίας Πλάμα. Μια προφορική τροπολογία. Κύριε Σέρκας. Δεν συμφωνούμε να ψηφίσουμε για την προφορική τροπολογία. Άρα την 24 υπέρ κατά αποχές. Η τροπολογία 24 στην αρχική της μορφή εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3.25 του κυρίου Κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 εστρέλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 ράπτη εστρέλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 μάκιντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 κα... υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, συμβιβαστική D. Από τέσσερις ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ε, παληθεύουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική D. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 26. Euh... Ε, Έχουμε 26 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται και οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Μετά από την παράγραφο 4, τροπολογία 34 της κυρίας Πλάμπ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 35, Εστρέλα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36, Μάκεταρ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος ε, συμβαστική ε. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Έγκρινεται μετά την παράγραφο 4 τροπολογία 38 Μάκινταρ υπέρ κατά αποχές. Έγκρινεται σε παράγραφος 5 τροπολογία 42 Μάνερ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43 της κυρίας Κόντς. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 μπεναμιάς είναι συμβατή ε, υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται αλλά υπαλληθεύουμε ηλεκτρονικά για την 39 Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας, 20 24, κατά, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 40 του κυρίου Μπουλόν ε, υπέρ, όχι, ναι, ναι, υπέρ. Κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41, μπιζότο, είναι συμβατή, την ψηφίζουμε. Με μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι. 41 λοιπόν όπως έχει τροποποιηθεί ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 41. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 5, συμβαστική F παρουσιάζεται από τέσσερις ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 της κυρίας Εστρέλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 6, 48 εσαγιά υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 48. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Τέλος της ψηφοφορίας. 23 κατά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 54. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49. Καταπίπτει. Les amendements 50, 51, 52, 53, 55 Οι 52, 53, 55 καταπίπτουν και μετά την παράγραφα 6 περνάμε στην τροπολογία 56 Ζουμπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 Πουπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 συμβαστική Ζ. Από τρεις ομάδες υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη συμβιβαστική G. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. «20 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται». Και φτάνουμε στην παράγραφο 7, στην τροπολογία 66 της κυρίας Ζούμπερ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνεται τα χέρια οπότε πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για 66 Tout le monde Le vote est clos. Ψηφίσατε όλοι.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 Λοιπόν, νομίζω πως έκανα μια ανοησία στην παράγραφο 6. Να πάμε λοιπόν λίγο πίσω για τις τροπολογίες 52 και 53, οι οποίες είναι συμβατές με την 54 την οποία εγκρίναμε προηγουμένως. Στη σύμφωνοι? Δεν ισχύει αυτό και για την 50, είπε κάποια. Donc nous allons voter le 50, 52, 53. 52 και 53 θα ψηφίσουμε. Ζητώ συγγνώμη και κυρίω, από όλους και κυρίως από τους συντάκτες των τροπολογιών γιατί βιάστηκα. Λοιπόν, πάμε πίσω και ψηφίζουμε γιατί στην παράγραφο 6 την τροπολογία 50 της κυρίας Ήρς πρώτα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Tout le monde a pu voter, 24 pour, 15. υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Και, και έτσι η 52 καταπίπτει, ενώ η 53 όχι και ψηφίζουμε για την 53 της κυρίας Στάινρουκ. Ποιοι είναι υπέρ της 53. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και γυρνάμε στην παράγραφο 7, μετά την παράγραφο 7, στην τροπολογία 67 της κυρίας Εντίτ Εστρέλα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, χωρίς τα λόγια που λέει if the female employment και τα λοιπά, μέχρι που λέει Ευρώπη, Στατηγική Ευρώπη 2020 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ α, της συμπερίληψης αυτών, αυτής της φράσης, υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Τέλος της ψηφοφορίας. C'est largement... Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7, 69 του κύριου Πουπάκη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 του κυρίου Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71, Κορνέλισεν και άλλοι, υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος. Tout le monde a bien voté, comme il voulait, bien suivi. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος ψηφοφορίας. 20 κατά, 24, συγγνώμη, 20 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Πάμε στην 72 του κυρίου Μπουλό με προφορική τροπολογία του ιδίου Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 72. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 73, ροντζούλη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74, πλάμ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75, της ιδίας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 8, συμβιβαστική AS Age. Αν θέλετε να επαληθεύσουμε την 75, να την επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, 36 υπέρ, 8 κατά. Όντως με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Λοιπόν, παράγραφος 8, συμβιβαστική AS Age, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, Επαληθεύουμε για την συμβαστική ΑΣ. Ε, Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 24 κατά απορρίπτεται. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες με τη σειρά 77. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 ράπτη και άλλοι υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται όντως. 78 καταπίπτει, 70... Όχι, δεν καταπίπτει, είναι συμβατή. Ε, την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 79 καταπίπτει. Η 80 καταπίπτει, 81 και αυτή. Όπως και οι 82 και 83. Και πάμε στην 84 μετά από την παραγωγή Ροντζούλη, υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται 85, έχει αποσυρθεί, παράγραφο 9, τροπολογία 86 Μάκενταρ που είναι ε, διαγραφής. Υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική EI από τέσσερις ομάδες, που είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην παράγραφο 10, στην τροπολογία 90 της κυρίας Τσίμερ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 μετά την τροπολογία... Συγγνώμη, 92, μετά την τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11, 93, μάκιντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 94 του κυρίου Μπέναμιας υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται 95. Αν θέλετε να επαληθεύσουμε, εντάξει, ε, άρχεται η ψηφοφορία για την 94. 94, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας, 26 υπέρ 18 κατά, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 95 είναι συμβατή, ψηφίζουμε του κυρίου Κάζα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 96 μετά την παράγραφο 11 τοπολογία 96 πλάμα υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται 97 εστρέλα υπέρ κατά. Αποχέ. να επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι. 26 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 98 ροντζούλη. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Τροπολογία 102 για διαγραφή υπέρ κατά απο, αποχές ε, απορρίπτεται ε, συμβιβαστική G από τέσσερις ομάδες πίνει είναι υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Στο εισαγωγικό τμήμα τροπολογία 108 Μάκιντάρ, η συγκίτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το σημείο α της παραγράφου 13, συμβαστική κάπα, από τέσσερις ομάδες που είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημείο Β, τροπολογία 114 Μακιντάριο για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 117 ε, μάλλον κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σημείο C 118 Μάκεντερ, η εισηγήτρια κατά υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 119 της εισηγήτριας, ποιοι είναι υπέρ, κατά Δεν σηκώνεται τα χέρια, οπότε θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλο le Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σημείο D. Συμβαστική L από τέσσερις ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, παλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. 21 υπέρ, 24 κατά. Δεν ε, απορρίπτεται. 120 της κυρίας Ήρς. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 121 καταπίπτει και το 122 και το 123. Πάμε λοιπόν στο σημείο ε, στην 124 της κυρίας Ρέγκνερ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές... Ηλεκτρονικός έλεγχος. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 20 pour, 25 contre, ça υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 125 μπιζότο, μπιτσότο, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 μάκινταρ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 13, μάλλον, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 128. Το μόνο monde Τέλος 30 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13. Με μεγάλη πλειοψηφία κιόλα. Παράγραφος 13, σημείο εα. Τροπολογία 127, χείριση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129, πλάμ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 13 σημείο ε, α νέο 130 της κυρίας Γκόντς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 της ιδίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 της ιδίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 3 της κυρίας Ήρση ποιοι υπέρ. Κατά Μα σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. 133. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Μάκιντάρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε την 137 της κυρίας Ροντσούλη με αίτημα για ψηφοφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα του κειμένου, χωρίς τις λέξεις rights and. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρα το δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα και ψηφίζουμε για την 138. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 εστρέλα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας 39 υπέρ 0 κατά 5 αποχές συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Et nous en revenons au point... Και φτάνουμε τώρα στο σημείο 10. Nous en, votons, nous en venons au point 11. Στο 11 μάλλον το σχέδιο δηλαδή του κυρίου Νταγντάν για την ενίσχυση τη οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρέ δυσκολίε να αφορά καν με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Το είπα. Θα ήθελα να ε, ε ψηφίσουμε για την πρόταση απόρρευση τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κυρίων Τσούμπερ και Λιαρίκ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Άρθρο 1, παράγραφος 2. Ε, Συμβαστική D. Από τρεις πολιτικές ομάδες. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, 47. Υπέρ παρακαλώ. Κατά Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, για την 47, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Για την 47. Πέρασε. 23 υπέρ 19 κατά 3 αποχές. Εγκρίνεται. 48. Φιλίπ Ντεμπάκερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 11 τώρα του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 49 της κυρίας Κορνέλισεν και Τούρουνεν. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε τριών πολιτικών ομάδων. Υπέρ παρακαλώ για τη συμβαστική ε. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα γίνει αμέσως ηλεκτρονική επαλήθευση. Tout Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 23 κατά ισοψηφία, άρα απορρίπτεται, αλλά άξιζε που το επαληθεύσαμε, δεν ήταν ε, προφανές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 12, το εισηγητή υπέρ, κατά, απόχες, ε, επαλήθευση για τη 12 παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ, ψήφισαν όλοι, πέρασε. 20 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν την 50 του κυρίου Μπουλόν σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, χωρίς το σε κάθε κράτος μέλος. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά, απόχες, εγκρίνεται. Ε, ποιος είναι υπέρ της προστήξης αυτών των λέξεων. Κατά, απόχες, Δεν θα προσθεθούν αυτές οι λέξεις. Τώρα θα ψηφίσουμε για την 51 του κυρίου Νταγντά, που συνάδει με την 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά άρθρο 3, παράγραφος 3, τροπολογία 13 του εισηγητή. Καταπίπτει. Και τώρα η τροπολογία 52 της κυρία Παπαδοπούλου με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 53 της ιδίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 54 για την παράγραφο 4 της κυρίας Κορνέλησεν και του υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 14 καταπίπτει και άρα πάμε στην ε, παράγραφο, 3 του άρθρου, παράγραφο 5 του άρθρου 3. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 55 του κυρίου Ντόιτσε που ανήκει σε μια ομάδα τροπολογιών. Έχουμε την 74, 77 και 80 μέσα στο ίδιο πακέτο. Συμβαστική νη και πι. Ε, ποιοι είναι υπέρ του πακέτου. Κατά. Αποχές. Η ομάδα 1 εγκρίνεται, άρα οι δύο καταπίπτει. Και τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε για το άρθρο 3 παράγραφος 6 τη συμβαστική Q από τέσσερις πολιτικές ομάδες ε, υπέρ της συμβαστικής κατά αποχές Εγκρίνεται αυτή η συμβαστική Q και περνούμε τώρα στην επόμενη συμβαστική F δηλαδή για το άρθρο 3 παράγραφος 6 σημείο α υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 3 έχουμε την ε, τροπολογία 63 κυρίας Κονέλησεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για το άρθρο 4, συμβαστική G, τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ. Τριών πολιτικών ομάδων, διορθώνει πρόεδρος. Green a ε, λέει. e δεν είναι η φιλελεύθερη, δεν είναι ALDE. Είναι η ίδια ομάδα. Εντάξει, τι φταίω εγώ που μπερδεύονται από μόνοι τους οι πράσινοι με τους φιλελεύθερους. Άρθρο 4, συμβαστική G, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, συμβαστική H, τριών πολιτικών ομάδων, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, ε, συμβαστική ΑΕ, δύο πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά άποχε. εγώ ισχυρίζομαι ότι απορρίπτεται. Με πιστεύετε, συμφωνείτε ή επαλήθευση. Απορρίπτεται, συμφωνείτε. L'amendement 67. 67 τώρα, Το εισηγητή υπέρ. Κατά Άποχες. Επαλήθευση. Για την 67 παρακαλώ. Μόνα a Πέρας. 17 υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται και άρα θα ψηφίσουμε τώρα για την τροπολογία 19 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στην 68 των κυρίων Κορνέλισεν και Τούρουνεν σε δύο τμήματα. Όχι, σε ένα τμήμα, διορθώνει ο Πρόεδρος, αλλά με προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση για την προφορική. Όχι, θα ψηφίσουμε για ολόκληρη την 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 69 του κυρίου Πριέτο υπέρ. Κατά. Άποχες Απορρίπτεται. Δεν τα πάτε πολύ καλά σε αυτό το άρθρο. 70. Ντεμπάκερ. Ζητάει χωριστή ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα, χωρίς το ε, όπου they were possible, επίπερ, κατά αποχές, εγκρίθηκε. Ε, και ποιος είναι υπέρ της προσθήκης τώρα. Κατά, ξανά, από την αρχή, υπέρ κατά αποχές δεν προστίθενται λοιπόν αυτές οι λέξεις, αποφασίστε. Και η 71 τώρα είναι συμβατή και άρα την ψηφίζουμε υπέρ της 71. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το άρθρο 6, παράγραφος 1 και φτάνουμε στην τροπολογία 72 υπέρ. Κατά αποχές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρθρο 6, παράγραφος 3, η 75, ίδια συντάκτρες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, η 20 του εισηγητή είναι συμβατή και την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα φτάνουμε στην 78. Κορνέλισεν και Τούρουνεν που είναι συμβατή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 6. Παράγραφος 5. Έχουμε ήδη ψηφίσει ε, την πρώτη ομάδα, τον μπλοκ 1, την έχουμε ήδη ψηφίσει, αυτή την τροπολογία, καλύπτοντας έτσι και τη συμβαστική Q. Και άρα για το άρθρο 9 μπορούμε να ψηφίσουμε για την τροπολογία 85, Κορνέλσιν και Τούρνεν πάλι, όχι. Και όμως... 85, Κορνέλης τούρνεν, ε, προτείνεται διαγραφή του άρθρου. Ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 10. Το νέο. Συμβαστική J. Δύο πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την 88 των Κορνέλισεν και Τούρνεν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 23 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα άρθρο 10, νέο πάλι. Συμβαστική ΚΑ, ΚΑΠΑ, από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα Άρθρο 11, παράγραφος 3, συμβαστική όμικρον, δύο πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα η 25 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 είναι συμβατή και άρα την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η άρθρο 11 παράγραφος 4 η συμβαστική π που καλύπτεται από την ομάδα 1, άρα δεν χρειάζεται και θα ψηφίσουμε για το άρθρο 12 παράγραφος 1 την 92 του κυρίου Ντεμπάκερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 92. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι οι πέρες. 24 είναι οι ψήφοι υπέρ 18 κατά και 4 αποχές. Εγκρίνεται 92. Και τώρα... Πάμε στα εκτιμώντα, στι αιτιολογικέ σκέψεις. Το 1, 27 του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 του εισηγητή καταπίπτει. Το ίδιο και 28 και άρα μετά το εκτιμώντας 1 φτάνουμε στη συμβαστική α τριών πολιτικών ομάδων υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας 1 πάμε στην τρία του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το Ε, 1 έχουμε την τροπολογία 29 της κυρίας Παπαδοπούλου με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 4 και 31 είναι ταυτόσιμε και θα τις ψηφίσουμε μαζί υπέρ. Κατά. απόχε. Εγκρίνονται. Κύριε Σέρκα, είστε κατά του εισηγητή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τροπολογία 32, ε, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές. Θα κάνουμε την απαλήθευση για την 32, παρακαλώ. Πέρας. 27 έναντι 19 ψήφων εγκρίνεται. Ε, τώρα η συμβαστική Β για το εκτιμώντας 2-3 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καταπίπτουν και φτάνουμε στη 35 του κυρίου Μπουλόν με νέο εκτιμώντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το, εκτιμώντας 3 συμβαστική λάμδα τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 καταπίπτει. Ε, τώρα στο εκτιμώντας 4 συμβαστική C2 πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα η 37 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 38 των Κορνέλσεν και Τούρουνεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 τώρα. Αυτή καταπίπτει. Και άρα πάμε στο εκτιμώντας 5 και ψηφίσουμε για την 39 των Κορνέλσεν και Τούρουνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, η 7 του εισηγητή καταπίπτει και φτάνουμε στο εκτιμώντας 6. Τροπολογία 8 του εισηγητή με μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Όχι, θα ψηφίσουμε τροποποιηθήσα 8 υπέρ. Κατά αποχές ε, θα γίνει επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι πέρας. 24 προς 18. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Et για τα εκτιμώντα 7 συμβαστική M τριών πολιτικών ομάδων ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Οι σοσιαλιστές ε, μου υπέδειξαν ότι υπάρχει ένα λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ψηφίσαμε τη 15 του εισηγητή page 3 de votre liste de vote. Στη σελίδα 3 του καταλόγου ψηφοφορία. l'article 3, paragraphe 5. Για το άρθρο 3, παράγραφος 5. Ε, Είχαμε ψηφίσει την ομάδα τροπολογιών 1, μπλοκ 1, η οποία όμως δεν κάλυπτα στην τροπολογία 15 που είναι συμβατή με τις 50 7 και 56. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είχαμε ψηφίσει και την 55 ή όχι. Όχι. Όχι, καλύπτεται η 56-57 περισσεύει μόνο του εισηγητή. Δέχεστε, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε για την 15 ε, του εισηγητή, παρακαλώ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία το σύνολο τη Έκθεση, Παρακαλώ. Είναι υπέρο ο παρόλε παρόλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν στο κείμενό του. Κλό. Πέρα. Εγκρίνεται η έκθεση με 36 ψήφου υπέρ, έναντι 6 κατά και 4 αποχών. Ε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Et ε, nous en Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 12 που είναι η ψήφιση της έκθεσης που συνδέεται με την προηγούμενη και επιγράφεται κοινέ διατάξει για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματο των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ. Είναι του κυρίου Ντόιτς. Υπάρχει μια τροπολογία παριθμών 16 της κυρίας Σούμπερ και του κυρίου Λεϊουαρίκε για απόρριψη του συνόλου της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ της 16. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 48 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε τη 49. Ψήφι υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Χρειάζεται επαλήθευση για το 49. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ψηφίσατε όλοι. 18 υπέρ, 25 κατά, δεν εγκρίνεται. Η τροπολογία 50 του κυρίου Νταρδέν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 51. Μπάκερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Άρθρο 3, παράγραφο 1, τροπολογία 8 του εισηγητή ψηφίπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Τη κυρία Πιτσότο είναι συμβατή υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. Άρθρο 3, παράγραφος 2, 53. Για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 54. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, τροπολογία 55. Κορνέλισεν και Τούρινεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ, 24 κατά, δύο εποχές. Ή 55 απορρίπτεται. Έτσι λοιπόν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 56 του κυρίου Χέλμετ. Ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 παράγραφος 1α 57 του κυρίου Ντεμπάκερ. Υπέρ. Abstention Κατά αποχές, 58 ε, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 59. Έχει αποσυρθεί. Α, δεν ήταν ε, παραδεκτή. 60 λοιπόν. Δεμπάκερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61. Που ζητεί απάλληψη υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 62. Μπιτσότο. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 66. Κονέλησεν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 καταπίπτει και τι ψηφίζουμε τώρα. 64 Κονέλισεν Τούρινεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 Νταρδέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 της κυρίας το ζητάει απάλληψη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 11 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 Μπιζότου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 μπουλά κατά αποχές εγκρίνεται 71 πισότο για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 της ιδίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 Κορνέλ Σεντούρινεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 Χέλμερ, συμβατή με την προηγούμενη πέ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 Το εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76. Μπορεί να ψηφιστεί, γιατί συνδέεται με την 73. Ψηφί υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, 77, τροπολογία Κορνέλη Σεντούζινεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε αυτό σας παρακαλώ. 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 17 υπέρ 26 κατά δεν εγκρίνεται, δηλαδή απορρίπτεται. 78 ντεμπάκερ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α6, ναι, παράγραφος 1α9. Ναι. Έχουμε τροπολογία 13 εισηγητή με προφορική τροπολογία. Διαφωνείτε με την προφορική. Όχι. Έτσι την ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ τη 13. Νο, νο, ποιος λέει όχι. Διαφωνείτε με την προφορική τροπολογία. Όχι. Ποιος είπε όχι. Ε, όχι ότι δεν έχουμε αντίρρηση. Δεν κατάλαβα. Το ΕΛΚ κάνει προφορική τροπολογία και ζητάει ε, να καταψηφιστεί. Καλά που κάνω και τη δουλειά του ΕΛΚ εγώ εδώ μέσα. Μήπως να μην τους ακούω καθόλου. Λοιπόν, το ΕΛΚ είναι κατά της προφορικής. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Αν συνέβαινε στους σοσιαλιστές μπορεί και να κάνω και το ίδιο. Ψηφίζουμε την αρχική 13. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79. Κορνέλισεν και Τούρινεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80. το υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81. Δαρντέν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 6 παράγραφος 4. Τροπολογία 82. Πίσω του υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Παράγραφ 4, 14. Την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83. Κορνέλισεν και λοιπά. Υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 83. Άρχεται η ψηφοφορία, Ψήφισετε όλοι, πέρας. 17 υπέρ, 24 ε, κατά, μάλλον δεν εγκρίνεται. Και με τις δύο εποχές πάλι δεν εγκρίνεται. Άρθρο 7, παράγραφος 1η, 84, τροπολογία πιζότο, ζητεί διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 7, παράγραφος 3. Υποπαράγραφος 1, 84 τροπολογια πιζοτο ζητει διαγραφη υπερ κατα εποχες απορριπτεται αρθρο 7 παραγραφος 3 υποπαραγραφος 1 συμβαστικη β από δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε έτσι στο άρθρο 7, παράγραφος 6, τροπολογία 88, πιζότο, υπέρ, ζητάει η διαγραφή κατά, αποχές απορρίπτεται, 89, Κορνέλη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8 παράγραφος 3, η τροπολογία 90 των ιδίων κυριών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 10α νέο, Συμβαστική σε από δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 του κυρίου Νταρδέν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 11 παράγραφο 1 υπό παράγραφος 2 νέα ναι. 92 Νταρδέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. άρθρο 11 νέο, συμβαστική D από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τώρα στο 12, μάλλον όχι ακόμα στο 12, παράγραφος 1, 96, πισώ του, ζήτη διαγραφή υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Και ερχόμαστε στην αιτιολογική σκέψη 1, 17, τροπολογία πισώ του, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Μετά 19 Κορνέλισεν Τούρνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 3, 20 μπουλών, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 21, πισω το υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 22, νταρδέν υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ιδεολογική σκέψη 3, 23, ντεμπάκερ είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 24, κορνέλισεν, τούρινεν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25, πίσω του υπέρ, καλά, κατά αποχές απορρίψεται. Οι δύο του εισηγητή είπε κατά αποχές εγκρίνεται. αλλά χρειάζεται έλεγχος γιατί δεν είμαι σίγουρη, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι τη δύο, πέρασε. 21 υπέρ, 20 κατά. Δύο εποχές δεν κρίνεται. Για την 28 τώρα δεν ξέρω ποια η μοίρα της. είναι συμβατή και μπορούμε να την ψηφίσουμε. 28 του κυρίου Πουπάκη, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 τόμα. Μαν, επίσης συμβατή, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 καταπίπτει. Ε, λογικη σκέψη σκέψη 6-29 της κυρίας Πισότο δεν ήταν ε, παραδεκτή. Η τρία του εισηγητού ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 30 της κυρίας Παπαδοπούλου ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 31 Το Μασμάν. συμβατή ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα 32 το απαράδεκτη. Η 4 του εισηγητή ψηφιπέ κατά αποχές Εγκρίνεται. 34 του κυρίου Πουπάκη. Συμβατή και την ψηφίζουμε. Ψήφι Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 33 του κυρίου Χέλμερ. Συμβατή. Ψήφι Π. Bien. Alors, l'amendement 33, qui est pour Contre 33 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 8. 36 Νταρδέν, Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 Το εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη. Έχει καταπέσει. Ζητώ συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Δικό μου λάθος. Ερχόμαστε λοιπόν στην 35 τροπολογία συμβατή με την 36 και την ψηφίζουμε ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 9, 6 του συγητή π. Κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά χρειάζεται μάλλον έλεγχος εδώ. Αρχίζει ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 17 υπέρ, 25 κατά, δεν εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 10, συμβιβαστική α, από δύο ομάδες υπέρ, κατά αποχές, η συμβιβαστική α εγκρίνεται. 11 αιτιολογική σκέψη, 41 του κυρίου που πάει και τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στην αιτιολογική σκέψη 12, 43 πισότο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42 Τόμας Μαν. Με ψηφοφορία κατά τμήματα που έχουν ζητήσει σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα χωρίς κάποιες λέξεις που βλέπετε εδώ. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Ποιο συμφωνεί με τις λέξεις που είχαμε βγάλει προηγουμένως. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε βγαίνουν αυτές οι λέξεις. Ε, η επτά καταπίπτει όπως και η... Έτσι δεν είναι. Α, όχι, 44 ψηφίζεται. Γιατί είναι συμβατή. Όχι, καταπίπτει και 44. Αιτιολογική σκέψη 13, 45. Κονέλη ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται 46 Νταρντέν συμβατή κατά αποχές εγκρίνεται 47 Χέλμε είπε. κατά αποχές απορρίπτεται και το σύνολο του κειμένου όπως αποποιήθηκε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που αρχίζει τώρα Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 36 υπέρ, 4 κατά, 3 εποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να συμπεριλάβουμε και τα κοινωνικά ζητήματα σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, τελειώσαν οι ψηφοφορίες και επιστρέφουμε στην Επιτροπή μας και ακριβώς την ώρα αρχίζουμε την ανταλλαγή απόψε με το Γενικό Εισηγητή για τον Προπολογισμό του 2013. Θα ήθελα να συνεχίσουμε. Σημείο 14. Euh, Ανταλλαγή απόψεων με τον Τζοβάνι ε, Λαβία που είναι ο Γενικός Εισηγητής για το Σχέδιο Προϋπολογισμού 2013. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαβία που ήρθατε. Για μας ε, έχει μεγάλη σημασία αυτή η ανταλλαγή απόψεων, διότι πραγματευόμαστε του γενικούς προσανατολισμούς του σχεδίου προπολογισμού για το 2013, καθώ και τις προτεραιότητες στον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης προετοιμάζεστε για τον τριμερή διάλογο που θα είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις ε, που θα γίνουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον προπολογισμό του 2013. Η γνωμοδότηση Επιτροπής Απασχόλησης Ενόψης του σε Διαλόγου θα προετοιμαστεί από τον κύριο Μπουλόν για το προπολογισμό του 2013 Ως εκ τούτου είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψε για το σχέδιο προϋπολογισμού. Ξέρω ότι κάθε επιτροπή έχει τις δικές προτεραιότητες και ότι πρέπει να πηγαίνετε σε όλους, αλλά τα δικά μας τα θέματα είναι ζωτική σημασίας. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεται να παρουσιάσω στην Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραμμές και την πορεία που θα ακολουθήσουμε για τον προϋπολογισμό του 2013. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός του 2013 είναι ο τελευταίος των δημοσιονομικών προοπτικών 2007 με 2013 και άρα είναι ένας προϋπολογισμός με τον οποίο θα ολοκληρωθούν πολλά από τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει την ίδια αυτή περίοδο. Και όπως όλοι οι προϋπολογισμοί, είναι ένας προϋπολογισμός ε, όπου θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ε, προτεραιότητες δράσης μας και να λάβουμε υπόψη και ποια ήταν τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει, ε, έχουν δηλαδή αναλυφθεί υποχρεώσεις τα προηγούμενα χρόνια και αναπόφευκτα θα πρέπει τώρα να γίνουν οι πληρωμές. Το θέμα των πληρωμών είναι το δυσκολότερο γιατί είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες περνούν μεγάλες δυσκολίες και δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η συμβολή πολλών ευρωπαϊκών χωρών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι μια συμβολή που κάνουν μέσα σε ένα πλαίσιο μεγάλων δυσκολιών και γι' αυτό το λόγο ήδη από πέρυσι τα κράτη-μέλη ε, τόσο στο Συμβούλιο και όσο και στη συνδιαλλαγή με το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό του προϋπολογισμού για το 2012 περιόρισαν εντόνως τις πιστώσεις πληρωμών και αυτό είναι ένα θέμα που θα επανέλθει και για τον προϋπολογισμό του 2013. Μόνο και μόνο για να σας δώσω ένα στοιχείο για να μπορέσετε να εκτιμήσετε την κατάσταση, θα σας πω ότι όσον αφορά την εκτέλεση του 2011, τα κράτη-μέλη ζήτησαν 15 δις ευρώ για τις πληρωμές μόνο το τελευταίο μήνα, το, το Δεκέμβριο. Αλλά η Κομισιόν μπόρεσε να πληρώσει μόνο ένα μικρό τμήμα αυτών, αυτού του κονδυλίου. 10 δις ευρώ που ήταν απαραίτητα για τη χρηματοδότηση του υποεκτέλεση προπολογισμού του 2011 μεταφέρθηκαν στις ανάγκες των πιστώσεων των πληρωμών του 2012. Και ήδη ο προπολογισμό του 2012 δεν ήταν και μεγάλο όσον αφορά τι πληρωμέ. Ήταν ένα προπολογισμό που προφανώ είχε ε, πόρου πολύ μικρότερου σε σχέση με τι ανάγκε. Αυτό μα οδηγεί στο... στο ότι το θέμα των πληρωμών αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ε, της δημοσιονομικής διαδικασίας και προφανώς μέσα στο 2013 θα πρέπει να το προσέξουμε όλους ιδιαίτερους και γι' αυτό ζητήσαμε να παρακολουθηθούν ε, ε, πολύ προσεκτικά οι πληρωμές από πλευρά Συμβουλίου και Κομισιόν, ώστε μέσα στον χρόνο να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης. Τώρα μόλις εγκρίναμε στην Ολομέλεια της περασμένης συνόδου τι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό και θελήσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μα σε δύο βασικά και μεγάλα θέματα που θα θέλαμε να αποτελέσουν τις κατευθυντήριε γραμμές για τον επόμενο προπολογισμό του 2013. Από τη μια πλευρά ανάπτυξη και ε, μεγέθυνση και από την άλλη το θέμα της απασχόλησης με ιδιαίτερη ε, αναφορά στην απασχόληση των νέων. η, τα ποσοστά ανεργίας ε, είναι τεράστια, ιδιαίτερα για τους νέους, ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα χρειαστούμε την προσπάθεια των ειδικευμένων επιτροπών για να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους λιγοστούς πόρους που έχουμε στη διαθέσή μας. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συναντηθούμε με όλες τις επιτροπές, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να εντοπίσουμε με τους ε, ε, συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στις διάφορες επιτροπές να εντοπίσουμε λοιπόν τις προτεραιότητες για το προπολογισμό του 2013. Πρέπει να εντοπίσουμε όχι μόνο θετικές προτεραιότητες δε, δηλαδή μίσο που προβλέπεται να υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών, αλλά θα πρέπει ε, επίσης να δούμε εάν υπάρχουν προγράμματα τα οποία υπολειτουργούν, που δεν χρησιμοποιούν πλήρως τα κονδύλια, ή προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι λιγότερο σημαντικά να προχωρήσουν, γιατί σε μια φάση κρίσης δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μόνο, τα, μόνο τις θετικές προτεραιότητες, αλλά να εντοπίσουμε και τις αρνητικές. Εκεί δηλαδή όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάποιους πόρους. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σαφές για το Ευρωκοινοβούλιο και είναι σημαντικό είναι το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί δεν διαφεύγει τη προσοχή σα ότι τα τελευταία 10 χρόνια το 85% των θέσεων απασχόληση δημιουργήθηκε από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν τη γραμμή ε, παρέμβαση λόγω των θετικών επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του στην απασχόληση. Ένα άλλο θέμα που παραδοσιακά είναι προσφυλές στο Κοινοβούλιο είναι το, τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα περιθώρια των εν λόγω κατηγοριών, δηλαδή ποια θα είναι τα κονδύλια που θα έχουμε στην διάθεσή μας για να χρηματοδοτηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα ανάλογο με αυτό του περασμένου χρόνου, με την έννοια ότι θέλουμε να υποβάλουμε καταρχήν τις προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις στην έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει την, ε, το κατά πόσο είναι σκόπιμο και, σκόπιμα και εφικτά. Για να μην μπλοκάρουμε χρήματα για πρωτοβουλίες που στη συνέχεια μπορεί να μην μπορούν να εκτελεστούν. Γι' αυτό ζητάμε από τις διάφορες, από τις διάφορες επιτροπές μέχρι τα τέλη του Μαΐου να ε, συγκεντρώσουν τις πρωτοβουλίες αυτές, δηλαδή πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικές δράσεις, που προτίθεται να παρουσιάσουν οι συνάδελφοι, ώστε μετά να στραφούμε στην Επιτροπή και εκείνη με τη σειρά της να κάνει μια αξιολόγηση σκοπιμότητας. Έτσι, στο τελικό πακέτο για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα που θα εγκρίνουμε, να συμπεριλάβουμε μόνο εκείνα τα προγράμματα που μπορεί να εφαρμοστούν. Να μην μπλοκάρουμε χρήματα για προγράμματα που μετά μπορεί να μην εφαρμοστούν. Κατά τα λοιπά, φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα. Να θυμίσω απλά ότι το επόμενο βήμα στην δημοσιονομική διαδικασία θα είναι η αξιολόγηση του Ευρωκοινοβουλίου επί τη βάση της ε, παρουσίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 25 Απριλίου του σχεδίου προϋπολογισμού. Αμέσως μετά λοιπόν θα αρχίσουμε στις όλες τις επιτροπές, τις κοινοβουλευτικές, τις δικές μας αξιολογήσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην εντολή για τον τριμερή διάλογο και τέλος στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού στα τέλη του έτους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση και για το ότι μας υπενθυμίσατε το πνεύμα του ψηφίσματος που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις γενικούς προσανατολισμούς για τον προϋπολογισμό του 2013. Για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εισηγητής είναι ο κύριος Φιλίπ Μπουλόν και ως εκ τούτου του δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαδία που είναι ο Γενικός Συγητής για τον προϋπολογισμό. Μας εξέθεσε τις προκλήσεις με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος ε, και κυρίως προκλήσεις, βασικότερες προκλήσεις για τον προϋπολογισμό το 2013. Πιστεύω ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, μια ευρωπαϊκή δυναμική, ούτως ώστε να εφαρμοστούν μέτρα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ε, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να τονίσω το ότι θα πρέπει μέσα από τον προπολογισμό 2013 να υποστηρίξουμε τους στόχους ε, της πολιτικής 2020 ε, και να χρηματοδοτήσουμε εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες όπως η νεολαία σε κίνηση, να χρηματοδοτήσουμε δράσεις όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην αγορά εργασίας είναι τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι και είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να βρούμε μέσα χρηματοδότησης για τις δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, χαιρετίζω την απόφαση να χρησιμοποιηθούν τα μία απορροφηθέντα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων, κυρίω σε σχέση με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, διότι ξέρουμε ότι εκείνε δίνουν την πλειοψηφία των νέων θέσεων απασχόλησης. Ε, Επαναπροσανατολισμό λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό θα τονιστεί δεόντω μέσα στο σχέδιο προπολογισμού 2013 και μέσα στο πλαίσιο του ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, Επίση, ζητείτε με μεγαλύτερη προσπάθεια σχετικά με την ανακύκλωση, επανακατάρτιση των κοινωνικών εταίρων για την εξέβρεση μισθωτών και για την ε, καλύτερη χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τονίζονται και τα προβλήματα που προκύπτουν ε, διότι ε, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση προτού εκταμιευθεί κάθε φορά ένα κονδύλι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το πρόβλημα και να το ρυθμίσουμε. Σε σχέση με την πρόσβαση στα όργανα μικροχρηματοδότησης και το πρόγραμμα EURES και το πιλωτικό πρόγραμμα για την εξέβρεση θέσει εργασία μέσω του Γιούρις. Όλα αυτά αναφέρονται μέσα στο σχέδιο προπολογισμού και το επικροτούμε. Θα θέλαμε να ξέρουμε η Επιτροπή Απασχόληση ε, ε, ποια, ποιο περιθώριο θα έχει σε σχέση με τα επιμέρου κονδύλια του προπολογισμού, αν θα μπορούσατε να μα ενημερώσετε το Eures, το Progress και η μικροχρηματοδότηση που υπάγονται στην κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, την ε, το κεφάλαιο αυτό δηλαδή του προϋπολογισμού και εφόσον υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καινοτομία θα μπορούσαμε μέσα από αυτή την έκθεση να τονίσουμε την ύπαρξη διαφόρων εμβληματικών πρωτοβουλειών που ευελπιστώ ότι θα χρηματοδοτηθούν το 2013. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω ότι φυσικά τα κράτη-μέλη θα έχουν το δικό τους ρόλο να διαδραματίσουν ούτως ώστε να αναλάβουν ρηξικέλευτες δράσεις που θα δημιουργήσουν θέσει θέσεις εργασίας. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό συντονιστικό ρόλο για να επιτύχει μια μεγαλύτερη κοινωνική σύγκληση και να δώσει μια αναπτυξιακή όθηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο επίτροπο Ανδόρ ε, είχε ανακοινώσει ότι τα αναπτυξιακά μέτρα και τα μέτρα στην αγορά εργασία θέλουμε να συμπεριληφθούν στο πακέτο τη οικονομική ε, διακυβέρνηση και τότε του απαντούσα εγώ ότι αυτό που ονειρεύομαι εγώ αντίθετα είναι μετά την οικονομική διακυβέρνηση να συσπηρωθούμε, να κινητοποιηθούμε ώστε να επιτύχουμε μια κοινωνική διακυβέρνηση μετά από την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, ε, κύριε Λάμπερτ, ευχαριστώ πολύ με την παρουσίασή σας. Και νομίζω ότι ε, έχετε μεγάλο δίκιο όχι μόνο για τις πιστώσεις πληρωμών και το ρόλο του Συμβουλίου εκεί, αλλά και τα υπόλοιπα που μας είπατε. Έχω μερικές ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτη ερώτηση. Εσείς πώς ορίζετε την αηφορία στην έκθεσή σας. Γιατί επαναλαμβάνεται ο όρος αηφόρος και δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς ευθυγραμμίζεται με την έννοια της αηφορίας, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή νέες τεχνολογίες πιο πράσινες, κατάρτιση, προσόντα, δεξιότητες, αυτό εννοείται. Ή μήπως μια βιωσιμότητα πιο μακροχρόνια και όχι αηφορία με την πράσινη έννοια. Επίσης, ξέρω ότι αυτό αγγίζει λίγο την επόμενη συζήτηση. Ε, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανεργία των νέων. Αλλά ένα από τα άλλα προβλήματα που έχουμε στην αγορά εργασίας είναι ακριβώς και το θέμα πώς ε, αυξάνεται η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης. Η ουσιαστική. Όχι τι θέλουν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί ο κόσμος όταν πατήσει τα 50 και είναι άνεργος είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρει δουλειά. Αυτό το σκέφτεστε ως ένα στοιχείο της στρατηγικής που προτείνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Άλλοι θέλουν το λόγο. Αν δεν θέλει κανείς άλλος, να πω κι εγώ ότι σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας ενώπιόν μας. θα πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι κλαδικές τομεακές προσεγγίσεις ε, σε σχέση με το ψήφισμα που εγκρίναμε, που ήταν γενικών προσανατολισμών μεν, αλλά κατανοώ ότι αυτό που σας ενδιαφέρει σας είναι η δημοσιονομική πτυχή. Εμείς από πλευράς της Επιτροπής μας, που είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως γνωρίζετε, ε, είδαμε στην τελευταία σύνοδο κορυφής μια μεγάλη διόρθωση να επανακινητοποιηθούν τα 82 δισεκατομμύρια του Ταμείου που δεν απορροφήθηκαν. Με την κλασική έννοια του προπολογισμού στα κράτη-μέλη, κανονικά θα έπρεπε να ψηφίσουμε ένα διορθωτικό προπολογισμό, έτσι δεν είναι. Εδώ δεν έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μετά αυτή την εξαγγελία από δημοσιονομική πλευρά συγκεκριμένα τώρα αυτό πώς θα λάβει σάρκα και όστα Γιατί το θέμα της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται διευκρίνηση. Πώς θα μεταφραστεί στην πράξη αυτή η εξαγγελία και ο προσανατολισμός και ποια θα είναι τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Διότι είναι ουσιαστικότατη η τροποποίηση του προϋπολογισμού και ως συνομοθέτες έχει σημασία μεγάλη να έχουμε σαφείς διευκρινήσεις. Για να μην πω να έχουμε και λόγο. Και ως Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει για τον προϋπολογισμό αυτόν τον διορθωτικό, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε και πώς θα εμπλακούμε. Γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε λόγια που δεν συνοδεύονται από έργα. Είχα το προνόμιο να δω το προσχέδιο και μιλήσατε για τις δεσμεύσεις των κρατών μελών και εξεπλάγει πολύ, εντυπωσιάστηκα. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε τι αντίκτυπο και επιπτώσεις θα έχει ακριβώς για την Επιτροπή μας. Αυτή η κινητοποίηση λοιπόν της τελευταίας στιγμής, τι σημαίνει, έχουμε καταλάβει πού αυτές οι πιστώσεις τελευταία στιγμής του παραπέντε πού θα πάνε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρατηρήσεις και τώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Ε, ξεκινώ με, από την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είχατε τη δυνατότητα να το δείτε. Ε, η πρόεδρος Μπερές ε, είδε πώς πάει η πώς προχωράνε τα αιτήματα τον τελευταίο μήνα κάθε χρόνο. Εδώ βλέπουμε ότι τον τελευταίο μήνα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτή η τόσο μεγάλη ζήτηση οδήγησε σε δύο αποτελέσματα. Από τη μια είδαμε ότι κάποια κρατημέλη δεν θέλουν να χάσουν λόγω του κανόνα νη συν δύο ορισμένους πόρους που προορίζονταν για τα ίδια. Οπότε είναι προφανές ότι μέχρι τελευταία μέρα, τελευταία στιγμή ε, έφερναν ε, λογαριασμούς προς εκαθάριση και υπήρχε ακριβώς αυτή η δέσμευση, κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία θέλησαν να αποφύγουν γιατί ήμασταν πίσω στις ε, ε, στα κονδύλια ε, ε, θέλησαν να αποφύγουν λοιπόν να χάσουν αυτά τα χρήματα, την απόλυτη των χρημάτων. Κάτι ακόμα που φάνηκε ήταν η αλλαγή του κανονισμού των διευθυντικών ταμείων που έφερε με ένα μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε κρίση. Και αυτή η αύξηση του τμήματος συγχρηματοδότηση οδήγησε ότι στο τέλο του χρόνου υπήρξε αύξηση τη ζήτηση και σε αυτά τα κράτη-μέλη. Ε, πρακτικά να σας πω ότι υπάρχουν χώρες που για την περιφερειακή πολιτική δεν ε, χρησιμοποίησαν 2,4 δις σε μια χώρα, δύο μια άλλη χώρα ε, και διάφορα εκατομμύρια κάποια άλλη. Δηλαδή εστιάζεται αυτή η δυσκολία πληρωμών σε κάποιες χώρες μόνο, κυρίως για προγράμματα τα οποία έχουν ε, υλοποιούνται μέσω του, των διαρθρωτικών ταμείων, του, του, του Ταμείου Συνοχής και κάποιοι προσπαθούν λοιπόν να ε, δώσουν προς εκαθάριση τους λογαριασμούς τους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και είδαμε ότι μέσα 2012 ποσά τα οποία προορίζονται σε άλλα προγράμματα θα, θα, θα έχουν δυσκολίες και ήδη προκύπτουν οι πρώτες δυσκολίες γιατί ήδη από χτες το τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για ορισμένες παρεμβάσεις με γελία ποσά, δηλαδή 18 εκατομμύρια ευρώ, όχι τεράστια ποσά, μέσα στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης αρχίζουμε να μιλάμε για την ανάγκη διορθωτικού προϋπολογισμού ενώ πρέπει να εκταμιεύσουμε όλα και όλα 18 εκατομμύρια ευρώ άλλα αιτήματα και βεβαίως σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα που υποβάλατε όπως σας είπα. Ε, είναι σωστό αυτό που είπε η συνάδελφος Λάμπερτ, ότι δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία. Το πρόβλημα είναι η ανεργία των ενηλίκων και στις κατευθυντήριες γραμμές μάλιστα εμείς μιλάμε για επίλυση, μπας περιπτώσει αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας εν γέννη. Και μετά προσθέτουμε με ιδιαίτερη ε, έμφαση στους νέους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλει στην άκρη και δεν θα λάβει υπόψη και τους υπολείπους ανέργους. Το θέμα είναι ε, αφορά τους, κυρίως τους ε, νέους αλλά και τους ε, ενήλικες που είναι ήδη σε κάποια προχωρημένη ηλικία και που χάνουν τη δουλειά τους και πολύ δυσκολεύονται να βρουν άλλοι. Τι σημαίνει Η φόρος θα πει τις ε, μακροπρόθεσμες πολιτικές. Ότι δηλαδή πρέπει να εφαρμόζουμε πολιτικές ή είδη παρέμβασης τα οποία να μπορούν να είναι βιώσιμα, αηφόρα. Αυτό σε όλους τους τομείς παρέμβασης. Αλληλεία, ας πούμε, αηφόρος, γεωργία, αηφόρος, που δεν μπορεί πια να είναι μόνο... Ε, οικονομικά αποδοτική ε, και για όλα τα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής και όλες τις άλλες πολιτικές ε, μιλάμε για αυτή την οριζόντια έννοια, την εγκάρσια έννοια της αηφορίας και σίγουρα η βοήθειά σας προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι πολύ χρήσιμη. Ο εισηγητής τώρα έρχομαι σε εσά τελευταία, γιατί, όχι γιατί είστε λιγότερο σημαντικό, αλλά σίγουρα γιατί θα έχουμε επαφέ στη διάρκεια τη δημοσιονομική διαδικασία. Θα έρθετε να συναντηθούμε, όπω είπα, και είναι σαφέ ότι πρέπει να διατηρήσουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών το λέμε ξεκάθαρα ότι σε αυτή το πνεύμα θα συνεχίσουμε. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι οι πόροι που υπάρχουν στον προπολογισμό συχνά δεν αρκούν για την επίτευξη αυτών των στόχων και το στο, νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει πιθανότατα να τροποποιήσουμε τη δομή των πολιτικών για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Στις προτεραιότητές μας έχουμε στηρίξει και φυσικά συμφωνώ μαζί σας ε, το τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το, ακριβώς λόγω του ρόλου που παίζουν για την καταπολέμηση της ανεργίας και κάνουμε και μια προσπάθεια για την επαγγελματική αλλαγή ή προσθήκη προσόντων γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους ε, εργαζόμενους αυτό. Επίση, συμφωνώ με τι προτεραιότητε που δίνονται στο Progress και τη μικροχρηματοδότηση. Είναι ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσβηλέ, δηλαδή η μείωση του χρόνου παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Κατάρτιση. Υπάρχουν ε, διάφορα προγράμματα τα οποία δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τι ανάγκε ε, ε, των προγραμμάτων ε, που προσπαθούν να βρουν νέα απασχόληση για όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω μετεγκατάστασης, λόγω παγκοσμιοποίησης. Έπειτα υπάρχουν και δισεκατομμύρια 82 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν είναι φρέσκα χρήματα, αλλά χρήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δεσμευθεί στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών. Και επίσης είναι εξίσου γνωστό ότι οι περιφερειακές πολιτικές είναι πολιτικές που ξεκινάνε από κάτω. Άρα οι προτεραιότητε ε, θα πρέπει να επιλεγούν από τις περιφερειακές αρχές που διαχειρίζονται τα προγράμματα. Και γι' αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό να ζητήσουμε από όλες τις διοικήσεις, τις περιφερειακές, να, να μετατρέψουν τα προγράμματα και να τα προσαρμόσουν με βάση αυτή τη διαθεσιμότητα που υπάρχει από πλευρά της Κομισιόν, όντως για να λυθεί το θέμα της ανεργίας, και αυτοί οι πόροι είναι σήμερα διαθέσιμοι και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Όμως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εντοπίσουμε και ε, πιστώσεις πληρωμών επαρκής για να μπορέσουμε να ελοπίσουμε τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω τις νέες τεχνολογίες. Α, δεν λειτουργεί. Θέλω να σας δείξω τη γραφιστική παράσταση. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα σας το μοιράσουμε αφού μας το έδωσε η συγητής, ε, για να λάβετε γνώση. Για αυτά τα 82 δις, αν κατάλαβα καλά, αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα γίνει απλώς μια συζήτηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, προβλέπεται πλέον να παρέμβει στην όλη συζήτηση. Ίσως δεν είμαι και παίων ε, για τα θέματα προϋπολογισμού, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή, ψηφίζουμε ένα σαν προϋπολογισμό, κατόπιν ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τροποποίηση της χρήσης των κονδυλίων αυτού του προϋπολογισμού. Αυτά τα 82 δις τι είναι, εν πάση περιπτώσει. είναι εξαγγελίες ή αντιστοιχούν σε κάτι από το ε, που ακολουθεί τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που υποστηρίχθηκε από το τελευταίο Συμβούλιο. Ε, ε, πείτε μας τι να λέμε. Μας λένε στις εκλογικές περιφέρειές μας έχετε κι άλλα τόσα δισεκατομμύρια καινούργια λεφτά. για να δούμε τι μπορούμε να τα κάνουμε. Πόσες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν με αυτά τα νέα δισεκατομμύρια. Θα προσπαθήσω να αποκαθαρίσω τι είναι αυτά τα 82 δις ευρώ. Όπως γνωρίζετε, οι πόροι των διορθωτικών ταμείων για την περιφερειακή πολιτική υποδιαιρείται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στο πλαίσιο των ε, κρατών μελών σε πολλές περιπτώσεις πάνε σε περιφερειακά προγράμματα. Η Κομισιόν έχει εγκρίνει λοιπόν αυτά τα προγράμματα και μετά από την έγκρισή τους ε, συνεχίζει και τα παρακολουθεί διαρκώς. Σήμερα λοιπόν μας λέει η Κομισιόν ότι 82 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχουν ακόμα δεσμευθεί και υπάρχει διάθεση της Κομισιόν να δεχθεί μια, έναν νέο προγραμματισμό για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Πρόκειται όμως για νέο προγραμματισμό στο πλαίσιο των λειτουργικών προγραμμάτων περιφερειακών, εθνικών, ανάμεσα στις ε, ε, αρχές της κρατικές και πάλι δηλαδή τα κάτι μελη θα πρέπει να τα διαχειριστούν αυτά τα χρήματα για μας αυτοί οι πόροι στο πλαίσιο της πολιτικής προπολογισμού έχουν προορισμό. Τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τον προορισμό τους, να τα μεταφέρουν από το ένα πρόγραμμα ή από, μια γραμμή παρέμβαση σε μια άλλη, άλλη γραμμή παρέμβασης. Η Κομισιόν λοιπόν ε, είπε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα και θέλει να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες εκ νέου προγραμματισμού των προγραμμάτων ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέε απαιτήσει επιχειρήσει που προέκυψαν στην περίοδο αυτή προγραμματισμού. Δεν πρόκειται όμω για φρέσκο χρήμα, γιατί μιλάμε πάντα για του ίδιου πόρου που περιλαμβάνονταν μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μιλάμε για νέε αποφάσει για τον προπολογισμό, γιατί για μα είναι πάντοτε χρήματα τη περιφερειακή πολιτική και άρα πάντοτε εκεί σε αυτέ τι γραμμέ βρίσκονται τα χρήματα αυτά. Άρα από την άποψη του προπολογισμού δεν θα αλλάξει τίποτα. θα αλλάξει όμως αν, κάτι αν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θελήσουν να αναπρογραμματίσουν τα όσα κάνουν ώστε να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για να λύσουν μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν ε, στην Ένωση. Σε ευχαριστούμε κύριε Ισηγητά αλλά διαπιστώνετε κι εσείς μια ουσιαστικότατη δυσκολία λόγω αυτού, διότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τα κράτη-μέλη συζήτησαν το θέμα επί μακρόν. Ε? Συζήτησαν για αυτά τα 82 δις σαν ήταν το α και το ω της αναπτυξιακής πολιτικής, πολιτικής πρόθεσης, ανταγωνιστικότητας, όλα τα κανάλια αυτά λέγανε και εξήγηλαν τα ανακαλά νέα. Όμως ουσιαστικά διαπιστώνουμε ένα φιάσκο, μια αποτυχία. Τα κράτη-μέλη δεν ε, χρησιμοποιούν χρηστά τα κονδύλια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή τους μέσω του προϋπολογισμού. Ε, εσείς μας μιλάτε για τον προϋπολογισμό του 2013, αλλά και για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα ισχύει αυτό. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτό. Τι επινόησε κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξήγηλε 82 καινούργια δις, ενώ δεν ισχύει τίποτα. Ορισμένε φορές ε, κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη και δεν απορροφούν ε, τα κονδύλια λόγω ζητημάτων συγχρηματοδότηση. Ε, δηλαδή, όσο λιγότερο απορροφούν τα κονδύλια, τόσο λιγότερη συγχρηματοδότηση έχουν να υπομισθούν. Λοιπόν, αυτά τώρα τα δίσε πρέπει να λειτουργήσουν ως κόδων κινδύνου και να πούμε ότι ε, ναι, ναι από τη μία δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα κονδύλια και από την άλλη όταν τα χρειαζόμαστε οι περιφέρειες ε, ε, δεν χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια ενώ τα χρειάζονται, δεν τα απορροφούν. Εν πάση περιπτώσει για τους επόμενους προϋπολογισμούς θα πρέπει να έχουμε αντλήσει τα εδάγματα και να μην επαναληφθεί αυτό. Τουλάχιστον η δική μας επιτροπή αυτή τι την κατεύθυνση θα ακολουθήσει σε κάθε περίπτωση επιτόπου ενδοϊπηρεσιακά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εξωτερικού συμβούλου. Οφείλουμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι για εσά. Η εισηγήτριά μα, κυρία Χάρκιν, είναι εδώ. Και Είπατε πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις για την ενεργοποίηση του Ταμείου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι για να ακολουθήσουμε ε, αυτή την στρατηγική θα πρέπει να πρικοδοτήσουμε αυτό το ταμείο μέσω ξεχωριστής γραμμής ε, στον προϋπολογισμό διότι έτσι ε, περιστέλλεται ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση των απορροφούμενων κονδυλίων αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό το θέμα σας απασχολεί στην Επιτροπή σας και τόσο άλλως θα έχουμε και μελλοντικά ευκαιρίες για να επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σιγητά για την επίσκεψή σας, για την ανταλλαγή απόψεων. Καλή δουλειά και να είστε σίγουρος ότι θα είναι θετική η γνωμοδότηση Επιτροπής Απασχόλησης ε, και για τις διαπραγματεύσεις εν του τριμερούς διαλόγου. Nous en avons terminé. Λοιπόν, και αυτό το σημείο και τώρα, σημείο 15 που συνδέεται με αυτό που μόλις ολοκληρώσαμε, ακρόαση. σχετικά με τις ευκαιρίες για τους νέους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους πολυάριθμους προσκεκλημένους μας. Η ιδέα της ακρόασης προέκυψε από την εξής απλή διαπίστωση. Με την έκθεση του Ρουνεν αναλάβαμε διάφορες πρωτοβουλίες Είχαμε ε, επίση την ε, ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίε για την νεολαία, πηχώντα ουσιαστικά τι εργασίε του Κοινοβουλίου και θελήσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε έναν απολογισμό να εξακριβώσουμε τι περιμένουμε ακόμη, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Ε, προς ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι το γνωρίζετε ήδη. Θα προσέθετα ότι πέρα από την ακρόαση έχει προβλεφθεί προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και ψήφισμα. Που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε προς έγκριση στην Ολομέλεια. Ποιοι είναι οι προσκεκλημένοι μας. Ε, Φραντσέσκα Μπαλτσάνη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είστε η γενική ε, εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του τρέχοντος το 2012 και άρα κάνετε ωραίο δίδυμο ε, με τον κύριο Λαβία για να μην υπάρξει διακοπή ανακολουθεί ανάμεσα στους δύο προϋπολογισμούς και γι' αυτό το λόγο θα σας δώσω το λόγο μετά τους ε, ε, προσκεκλημένους. Ο ε, κ. Δεπού που είναι εκπρόσωπος της Γενικής Διεθνής Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολείται με το θέμα της πρωτοβουλίας για τις ευκαιρίες για τους νέους. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία που εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής 2020. Παρακαλώ, έχει τη διάθεσή 8 ως 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ήταν όχι μόνο να σας παρουσιάσω την πρωτοβουλία την οποία πλέον καλώς γνωρίζει και η Επιτροπή σας αλλά για να σας ενημερώσω καλύτερα για την κατάσταση των εργασιών που προβλέπονται για την υλοποίηση. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν όπως γνωρίζετε εξεγγέλθη από τον Πρόεδρο Μπαρόσο στην ομιλία του στο Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την καταθέσαμε το Δεκέμβριο δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι ανταποκρίνεται σε μια πολιτική όσο και κοινωνική επίγουσα ανάγκη διότι βλέπουμε να αυξάνεται η ενεργεία των νέων με τρόπο ε, ανισχυτικό και ανώμαλο ε, με ρυθμούς που έχουν πολύ ανισχυτικά ποιοτικά στοιχεία διότι συνδέεται με μεγάλη αύξηση το ποσοστό των νέων που είναι εκτός της εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης και εκτός εργασίας. Και παγιώνεται επίσης αυτή η ανεργία. Έχουμε νέους μακροχρονίους άνεργους πλέον, όλο και περισσότερους, ε, μεταξύ της ηλικιακή ομάδας των νέων ανέργων. Αυτή η εξαγγελία λοιπόν του Προέδρου Μπαρός ακολουθήθηκε από την παρουσίαση της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέλη Δεκεμβρίου όπως σας είπα και εσείς ήδη τονίσατε κυρία Πρόεδρε ότι ε, γνώρισε μεγάλη απήχηση στην άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου. Αυτή η πρωτοβουλία είχε σαφή στόχο τη λήψη κάποιων μέτρων για να δρομολογηθούν επίγουσες ε, ενέργειες για κάποια ειδικά προβλήματα. Βεβαίως το, ζήτημα της απασχόλησης γενικότερα εγγράφεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Θα επανέλθουμε σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επανέλθει με την παρουσίαση κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου αυτού που σήμερα πλέον ονομάζεται ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Θα είναι μια ανακοίνωση και έγγραφα εργασίας που θα ασχολούνται με την εργασιακή πολιτική ευρύτερα, γενικότερα σε ένα ολόκληρο πλαίσιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται η σημερινή ανακοίνωση που ε, κάπως ε, προηγήθηκε γιατί είναι και προτεραιότητα η εργασία των νέων. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή έχει τέσσερις ε, τομείς προτεραιότητας εντοπίσει. Ε, όλο και περισσότερο αυξάνεται η πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου και θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό. Είναι μία ενότητα. Δεύτερη ενότητα να αντιστοιχούν οι νέοι στις ανάγκες αγοράς εργασίας ως προς την εκπαίδευσή τους. Τρίτη ενότητα ε, να υπάρχει σωστή προσφορά ε, κατάρτιση στους επαγγελματικούς χώρους, on the job training λέγεται αυτό στα αγγλικά, με διάφορες μορφές τις οποίες θα επανέλθω στη συνέχεια και γενικότερα η διευκόλυνση ε, της πρόσβασης σε μια πρώτη θέση εργασίας. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία έχει και δύο πτυχές εκτός από τα τέσσερα σκέλη. Η πρώτη πτυχή, η βασική, ε, ε, απευθυνόταν στα κράτη-μέλη που είναι καθήλυνα αρμόδια. Και η δεύτερη σε κάποιες πρωτοβουλίες ειδικέ και συγκεκριμένες που αναλογούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει κάποιων δημοσιονομικών δυνατοτήτων που είχε για το οικονομικό έτος του 2012 αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα κρατημέλη, η πρόθεσή μας αφήσει ήταν να, κάνουμε, να αρχίσουμε ένα πολιτικό διάλογο με τα κρατημέλη, γιατί ε, στατιστικά ε, σε εκείνες τις χώρες που έχουν περισσότερη ενεργεία των νέων για να ε, αναπτύξουν ατζέντε, προγράμματα εθνικής δράσης, έτσι ώστε να φτάσουν καλύτερα στους στόχους ή να ακολουθήσουν τις προτεραιότητες της ανακοίνωσης. Και ένα που άκουσα τελευταίο που συζητούσατε προηγουμένως, κάνοντας καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπάρχουν στη διάθεσή τους, είτε είναι αυτό το κοινωνικό ταμείο, είτε πόροι και πιστώσεις από τα ταμεία συνοχής. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν αυτή η δράση, η πτυχή της ε, ανακοίνωσης έλαβε μια διτή μορφή. Ομάδες δράσης αφενός, τα 8 κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή έχουν την υψηλότερη ενέργεια των νέων και από την άλλη μια σειρά συσκέψεων, έτσι, διμερών στις Βρυξέλλες με τις εκάστοτε αντιπροσωπείες, τις μόνιμες, των 7 άλλων κρατών μελών που εκτός από τις 8 πρώτες έχουν εξίσου αυξημένη ανεργία στους νέους σε σχέση με το μέσο όρο. Πάντα ήταν ε, πολιτικός ο διάλογος και εγκάρσιος ε, εκπροσωπούντο ε, πολλές γενικές διευθύνσεις και η περιφερειακή και η οικονομική και η γενική διεύθυνση των νέων και διπλή λοιπόν αυτή η διάσταση και πολιτική Λοιπόν, αυτές οι διμερείς οι σκέψεις ήταν μία μόνο φάση σε μία ολόκληρη διαδικασία. Γιατί δεν είναι άπαξ αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να είναι διαρκής και μόνιμη η επαφή και η συνεργασία με την εκάστοτε αντιπροσωπεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης θα κάνουμε από την Επιτροπή και μία έκθεση στα ε, μέσα της περίοδου. Έγγραφο εργασία λοιπόν των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπή θα ανακοινωθεί και θα είναι στοιχείο του πακέτου για την απασχόληση και βεβαίω θα ενημερωθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλος ιδιαίτερος η Επιτροπή σα. Αλλά παρακαλώ κρατήστε το, είναι διάμεσο αυτό το έγγραφο, δεν είναι τελικό, είναι στα μέσα τη περίοδου, είναι προσωρινό απορρέει από τις επαφές με τα κράτη-μέλη και θα δώσει μια πρώτη ένδειξη για την κατάσταση των πραγμάτων. Και τι κάνουν τα κράτη, πώς προγραμματίζουν ή πώς ε, αναπρογραμματίζουν ε, και αν διοχετεύουν ε, κάποιους αναπορόφητους πόρους από το Κοινωνικό Ταμείο με νέα σχέδια, έργα και πρωτοβουλίες υπέρ της επασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη μετεκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη μάθηση και την προσφορά περίοδων άσκησης. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υλοποιήσει μια σειρά πρωτοβουλειών το πλαίσιο ποιότητας για τις ε, περιόδους άσκησης, τα λεγόμενα στάζ, ήταν ένα έντονο αίτημα ε, των ε, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των νέων στην Ευρώπη και θεμητό. Θα γίνει και διαβούλευση, ε, είναι ένα στοιχείο του πακέτου αυτού για την απασχόληση και θα μας επιτρέψει κανονικά να έχουμε τα αποτελέσματα ταυτόχρονα με μια μελέτη που μόλις δημοσιεύσαμε για να λάβουμε μια πολιτική πρωτοβουλία με συστάσεις πριν τα τέλη του έτους. Εγγύησεις για την απασχόληση υπέρ των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πραγματικά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και ο Πρόεδρος της πάρα πολύ και το υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο που μας ζήτησε να ε, ε, ετοιμάσουμε μια προκαταρκτική δράση. Mm. Για να υλοποιηθεί λοιπόν αυτή και αν όλα πάνε καλά θα μπορέσουμε να εξαγαγούμε τα απαραίτητα πολιτικά διδάγματα για να εκπονήσουμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ίσως και το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η σύσταση αυτή πριν τα τέλη του έτους. Μίλησα για τη μαθητεία προηγουμένως. Ε, είναι σαφές ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσουν. Χαιρόμαστε και ξέρω ότι ο Πατρίκ Λτσέτ και ο Μαξίμ ξέρω ότι θα μιλήσουν αργότερα. Ε, χαιρόμαστε για τις ε, πρωτοβουλίες και της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ή κάθε μια οργάνωση από την πλευρά της για να κάνουν αυτά που της αναλογεί, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίως θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. απελευθερώνοντας κονδύλια για τεχνική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε και να βοηθήσουμε για προγράμματα μετάβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση στα κράτη-μέλη με περιόδους μαθητείας και άσκησης για να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων. Και ταυτόχρονα τελειώνω ε, λέγοντας ότι θα υποστηρίζουμε και τους νέους ε, για να έχουν πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα με κονδύλια για τεχνική υποστήριξη και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της τάξης των 3 εκατομμυρίων για να μπορέσουν να υποστηριχθούν κάποια σχέδια στα κράτη-μέλη για τους νέους επιχειρηματίες επιπλέον βεβαίως των όσων ήδη γίνονται από το μέσο της μικροχρηματοδότησης, αυτή τη διευκόλυνση που γνωρίζετε. Όλες αυτές λοιπόν οι πρωτοβουλίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ λειτουργική διάσταση σε αυτή την προσπάθεια. Η διάμεση προσωρινή έκθεση θα διαβιβαστεί και στο Συμβούλιο και βεβαίως στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου και προβλέπεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια συνολική έκθεση για την υλοποίηση και παρουσίαση αυτής στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Και βεβαίως κανονικά κυρία Πρόεδρε θα είναι στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή σας ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Euh, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, γενική εισήγηση και ερχόμαστε στους τέσσερις προσκεκλημένους μας. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στην κυρία Florence Μοριγιόν από την Ένωση Επισφαλής Γενεά.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 Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια στοιχεία κλειδιά για να δείτε ποια είναι η δύσκολη κατάσταση των ε, νέων. Στο 2006 ζητούσαν 800.000 ε, σταζιέρ στην Γαλλία, ενώ σήμερα ε, είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία. Η σταζιέρ είναι μια πραγματική βιομηχανία. Είναι δηλαδή μια εφεδρεία σε φάση κρίσης που επιδεινώνει την τη δυσκολία της ανέβρεσης ε, θέσης απασχόλησης. Αυτή η επισφάλεια που γενικεύεται βαραίνει όσον αφορά τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις για τους μισθούς. Ε, οι μισθοί έχουν μετιμειωθεί 10% τα τελευταία χρόνια. 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα ΑΕΠ μισού δις πρόκειται για 200 εκατομμύρια ευρώ που πάνε στο κεφάλαιο ενώ οι εργαζόμενοι αναζητούν την ισορροπία. Ε, ναι. Κάποιος διακόπτει την ομιλήτρια γιατί δεν γίνεται να μεταφραστεί με την ταχύτητα που διαβάζει. 200 δις ε, σημαίνει δύο φορές ε, τον ε, προϋπολογισμό για την, εθνικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Θα μπορούσαμε να πούμε για μηχανισμούς ελέγχου, την πολιτική θητεία, τα στάζ. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε ένα συμπλήρωμα συνεισφορών των επιχειρήσεων όπου η, ο αριθμός των επισφαλών θέσεων απασχόλησης είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο. Θα μπορούσαμε επίσης να συστήσουμε να περάσουμε στην εβδομάδα των τεσσάρων ημερών, σύστημα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στη Γερμανία. Ε, αυτό θα σήμαινε βελτίωση, μείωση μάλλον του χρόνου εργασίας στην κατά μέσο όρο 20% καθώς και την ε, μείωση του, του φόρτου. Στη Γαλλία θα σήμαινε αυτό ένα 1,5 έως και 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης επιπλέον. Γιατί η ανεργία είναι αντιπαραγωγική και μακροπρόθεσμα. Καθώς και τα στάζ, το να πιέζεται πολύ το εργατικό δυναμικό ε, είναι αντιπαραγωγικό. Για παράδειγμα, στη δική μου ηλικία η μητέρα μου είχε, ήταν δύο φορές ιδιοκτήτρια και είχε και τρία παιδιά. Ήταν ιδιοκτήτρια δύο περιουσιακών στοιχείων δηλαδή ενώ ε, όπως και πολλοί νέοι ε, σήμερα και εγώ ονειρεύομαι μια σταθερή δουλειά και ε, κάποιο κατοικία. Πολλοί νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ένα παιδί. Α, πόσο μάλλον να μιλήσουμε για το μέλλον, γιατί διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στους ε, άνεργους και την μάζα εκείνων που προσωρινά απασχολούνται. Αυτό δεν πρόκειται να επιταχύνει την ε, ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη είναι αυταπάτη ούτως ή άλλως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά εκλογικά προγράμματα και η Ένωσή μας έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα για να επηρεάσει τα πολιτικά κόμματα που ονομάζεται Young and Poor, νέοι και φτωχοί δηλαδή, ε, και προσπαθούμε να επηρεάσουμε τα πολιτικά κόμματα, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 2,2% την περίοδο 80 με 89, 1,2% μέχρι το 99 και 1% για την περίοδο 2000 με 2009. Επίσης πλέον δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την βεβαιότητα μιας επάπειρων ανάπτυξης σε έναν ε, πεπερασμένο πλανήτη. Ε, είδαμε ότι υπάρχει μείωση της ε, παραγωγής πετρελαίου το 2006 και από τότε και μετά δεν πάβει να αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Πρέπει να ανάξουμε λοιπόν τα πρότυπα ανάπτυξης εάν δεν θέλουμε να ξεφύγει από τον έλεγχό μας η κατάσταση του πλανήτη. Επίσης ε, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να αναστραφεί αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα μαζικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελούν και ένα μέγα κοίτασμα νέων θέσεων απασχόλησης. Ε, επενδύσεις στην οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας και στην, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 2000 με 2009 ήταν η πιο ζεστή περίοδος που είχε καταγραφεί και το 2010 ήταν το πιο ζεστό έτος που είχε ποτέ καταγραφεί σύμφωνα με την NASA. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το όριο των, του 2% αύξησης αύξηση της θερμοκρασίας, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στην μετακίνηση 200 εκατομμυρίων ανθρώπων και άρα και σε μεγάλες συγκρούσεις. Θα πρέπει να αυτό να προβληθεί για να μην διαπιστώσουμε την ε, κατάρρευση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαστήρι. Ποιον, Ποιον ωφελεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Και τέλος θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την κατάσταση της, ε, που μοιάζει με την Ρώμη. Ε, η Ρώμη φτιάχτηκε από διάφορους ε, λαούς, η τεχνολογία τους ήταν, μάλλον υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων που ήξεραν μόνο να αγωνίζονται, να πολεμών. Δεν έκαναν ποτέ διαφοροποίηση απέναντι στους διάφορους βάρβαρους που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Σας ευχαριστώ. Ήταν σαφέστατο και ηχηρότατο το μήνυμά σας ε, για την ε, να υπομιστούμε όλες τις ευθύνε μας από το Φόρουμ Νεότητας ε, τώρα Τζουζέπε Πορκάρο. Ευχαριστώ. Θα παλαιαμιλήσω αγγλικά. Thanks for the opportunity. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας παρακολουθεί και δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό για την αντιμετώπιση της κρίσης ε, της νεολαίας από τα τέλη του 2008 όταν το πρώτο σοκ, νιώσαμε το πρώτο οικονομικό σοκ. Αυτά που έχουμε παρατηρήσει και καταγράψει όπως μόλις είπε και η συνάδελφός μου, είναι η επιδείνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι νέοι. Όλο ένα και περισσότερο. Τώρα, επιτέλους, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο των θεσμικών οργάνων αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα. Πρώτη φορά έγραψε στην μερίσια διάταξή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Ξέρουν ότι δεν είναι πλέον βιώσιμη η κατάσταση. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι έπρεπε να περιμένουμε να χειροτερέψουν τόσο τα πράγματα ώστε ε, το είπα το όργανο λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει να ε, εξετάσει και να ρυθμίσει το ζήτημα. Ένα από τα βασικά θέματα ως προς την προσέγγιση μας ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι το εξής. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το πρότυπο για να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε και τις επιπτώσεις ε, της κρίσης. Βλέπουμε ότι τα μέτρα λιτότητας ε, δεν θα αρκέσουν. Το έχουμε συνειδητοποιήσει και χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, αναθεώρηση του αναπτυξιακού μοντέλου με ενοποιημένο τρόπο, τόσο ώστε η πολιτική απασχόληση, η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική ανταγωνιστικότητα ε, όλες αυτές οι πολιτικές ε, να συνδυαστούν και σε αυτό οι νέοι διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Σε σχέση συγκεκριμένα με αυτή την πρωτοβουλία για τους νέους, πρόκειται για το θέμα που συζητούσατε προλίγου, δηλαδή δεν ε, υπάρχουν φρέσκα λεφτά δεν είναι αυτό το θέμα. Ούτε καν ανακατανομή των ε, σταμένων κοντιλίων δεν προβλέπεται. Ε, αναπρογραμματισμός, πιθανός αναπρογραμματισμός των εφιστάμενων πόρων. Αυτό είναι το θέμα μας. Εάν λοιπόν θεωρείται τόσο σημαντικό το θέμα των νέων που ανακάγεται σε προτεραιότητα, μας ξαφνιάζει που η μόνη λύση στην οποία καταλήξαμε είναι ο αναπρογραμματισμός και ούτε καν εφαρμογή του αναπρογραμματισμού γιατί είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Ε, παραμένουν όλα ομιχλώδη και ασαφή ως προς την εκτέλεση. Οπότε δεν ανησυχούμε για αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν σε εθνικό επίπεδο. Ως προς την ίδια την υλοποίηση, θα κάνω και μία τρίτη παρατήρηση. Υπάρχει ανεξερεύνητο δυναμικό σε σχέση με τα προγράμματα που προτείνονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τους νέους ε, σε συνεργασία με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών όχι μόνο έχουμε εκπληκτική σχέση με τους νέους, αλλά και ουσιαστική τεχνογνωσία που συμμετέχουν, συμβάλλουν και οι ίδιοι οι νέοι στις δράσεις και γι' αυτό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Θερμή έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να διευκολύνει αυτή τη συνεργασία και την πρόσβαση στην χρηματοδότηση που συζητείται τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί η κατάσταση των νέων επίσης ένα συγκεκριμένο κονδύλι να διοχετευτεί ακριβώς για τις οργανώσεις των νέων. Ένα κομμάτι θα προέρχεται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς όπως για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στη Φινλανδία ε, αλλά πρέπει να προωθήσουμε την ε, ενεργό ηθαγένεια καθώς και την δράση των οργανώσεων των νέων. Τέταρτο και τελευταίο σημείο οι μαθητείες ε, στα πλαίσια επιχειρήσεων είναι ένα σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αλλά όπως είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ σε συνεργασία με ε, την ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και συγκεκριμένα οργανώσεις για τους ε, νέους και σε συνεργασία με βουλευτές του Κοινοβουλίου όπως η Έμιλη Τωρινή προωθούμε τις μαθητείες αλλά υψηλών δεξιοτήτων. Σας παραπέμπω και στο Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις μαθητείες θα ήθελα να ε, προσυπογραφεί από όλου και στις 16 Μαΐου θα έχετε τη δυνατότητα συγκεκριμένα έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα γίνει παρουσίαση από κοινού με τον Πρόεδρο Σούλτς. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε από πλευράς των συνδικάτων ο κύριος Πατρίκ Ιτσέρ που είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΤΟΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία ε, να <clears throat> καταθέσουμε τη μαρτυρία μας σήμερα. Κανονικά οι νέοι θα έπρεπε να είναι το μέλλον μας, να εκπροσωπούν το μέλλον μας. Και σήμερα ξέρουμε ότι είναι από τις πιο ευάλωτες ε, ε, ομάδες. Είναι η παράμετρος προσαρμογής στην κρίση και με την ανεργία, με την επισφάλεια, την ανασφάλεια, όλο και περισσότερες μαθητείες στάζ με ε, αποτέλεσμα δημογραφικά προβλήματα και ακόμα και συνδικαλιστικά ε, αναγκάζονται να, να συγκατοικούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν ε, είναι ανεξάρτητοι οικονομικά. Υπάρχει μια πρωτοβουλία για τις ευκαιρίες των νέων. Δεν αμφιβάλλω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με αυτό, αλλά είπατε κι εσείς οι ίδια ότι όλα αυτά είναι εξαγγελίες. 30 με 82 δισεκατομμύρια και ξέρουμε ότι οι πόροι αυτοί ούτε θα ε, διατεθούν, ούτε θα δαπανηθούν. Πώς λοιπόν, να σκεφτεί κανείς ε, ότι μετά τη task force που έχει πάει στην Αθήνα θα μπορέσει η Ελλάδα να συγχρηματοδοτήσει κάτι σοβαρό για τους νέους. Και βεβαίω θα επιστρέψουν τα χρήματα προς τα κράτη-μέλη διότι δεν θα απορροφηθούν. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Είναι ημίμετρα κάτι εκατομμυριάκια. Ε, κατά τα άλλα, ε, θα πρέπει να ε, αναρωτηθούμε αυτές οι ομάδες δράσης, οι task force, τι θα πάνε να λένε στις κυβερνήσεις. Πέρα από την ενδιάμεση έκθεση θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν και μάλιστα οι νέοι. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε να πιστεύουν ότι να, να, να προσποιούμαστε ότι θα λυθούν τα προβλήματα με την ευελιξία, με μισθούς πείνας, η πρόσληψη των νέων, αυτά κρύβουν το πρόβλημα και το μεταθέτουν. Θα φέρουμε αντιμέτωπες ομάδες ε, ηλικιακές και εργαζομένων ε, με ανέργους ε, απέναντι. Και αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βυθίζουν κάποιες χώρες όπως και η Ελλάδα στην ύφεση. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η πίτα της απασχόλησης με θέσεις εργασίας ποιοτικέ, ένα new deal ουσιαστικό, σχέδιο επενδύσεων, ε, όχι μόνο για τις επενδύσεις ε, και την ανάπτυξη αλλά και για τις θέσεις απασχόλησης γιατί υπάρχει και η άνεργη ανάπτυξη. Και ε, βεβαίως ε, χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ε, είναι σε δυσκολία, οπότε χρειάζονται ευρωομόλογα, φόρους επί των χρωματοοικονομικών συναλλαγών κτλ. Θα πρέπει να έχουμε το, το παράδειγμα στο παρελθόν είχαμε τη Δανία, σήμερα τη Γερμανία. Αν είδε η Γερμανία το 2010 να αυξάνεται κατά 8% τις ε, εξαγωγές, το 1% μόνο είναι η συγκράτηση των μισθών και το 7% είναι καινοτομία, έρευνα, κατάρτιση των εργαζομένων κτλ. Μιλούν σήμερα οι ηγέτες μας, οι πολιτικοί για ανταγωνιστικότητα και μας λέγουν ότι υπολοιπόμεθα της Κίνας και της Ινδίας. Άρα μειώστε 30% τους μισθούς στην Ελλάδα. Και κυρία Πρόεδρε, θα σας παραθέσω, εσείς είπατε σε κάποια άλλη ακρόαση ότι το, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσουν να θέλουν να κάνουν τους Ευρωπαίους Κινέζους. Ε, ε, ποιοτική λύση χρειάζεται προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω και για την Ελλάδα, με επενδύσεις. Πολύ σύντομα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων βεβαίως υποστηρίζει τη Youth Guarantee, την πρωτοβουλία αυτή, όπως και το χάρτη που προτείνει το Φόρουμ των Νέων όλα αυτά που λέγονται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εγκατάλειψη του σχολείου, ε, το διπλό σύστημα μαθητείας και σχολείου, όλα αυτά είναι καλά. Θυμίζω ότι το 2010 κοινωνική κοινωνικοί εταίροι ε, ε, υπέγραψα μια συμφωνία για την αγορά εργασίας και για τους νέους. Θα τα πει ο Μαξίμ, τα είπε και ο κύριος Δεμπάουερ προηγουμένως. Και εμείς ως κοινωνική εταίρη καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα πρόγραμμα εργασίας 2012-2014 των κοινωνικών εταίρων, όπου η ανεργία γενικώ και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων είναι προτεραιότητα. Η καταπολέμηση της προφανώς. Στον τριμερή κοινωνικό διάλογο τα συζητήσαμε αυτά και ελπίζω ε, η διάσταση αυτή των νέων να αρχίσει να ε, υλοποιείται από τον Ιούνιο, γιατί οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να βοηθήσουν, το είδαμε σε πολλά κρατημέλη και στη Γαλλία, με τη συνοδεία, την πλαισίωση των νέων ε, για τη στέγασή τους, πολέμηση ε, των υπερβολικών καταχρήσεων στα στάζ, ένα ε, θέμα επιθεώρησης εργασίας, συγκεκριμένες προθεσμίες που θα πρέπει να τηρούνται ανάμεσα σε δύο μαθητές και ως Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων θα πρέπει και εμείς να έχουμε προτάσεις, υπεύθυνα μέτρα και δράσεις και πρέπει να πω ότι στο τελευταίο συνέδριο στην Αθήνα ε, η Επιτροπή των Νέων μας ε, απέκτησε δικαίωμα ψήφου. Έχει λοιπόν πλήρη λόγο και ψήφο, συμμετείχε στην κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, συμμετείχε στο κοινωνικό διάλογο, το τριμερί τους ε, ζητήσαμε να αξιολογήσουν την πρωτοβουλία για τις ευκαιρίες των νέων και βεβαίως μαζί με τους νέους μας θα κάνουμε την εκστρατεία Είδατε τη με το Φεβρουάριο που ε, λέγεται αυτή η πρωτοβουλία τχόσετρο, ε, φτάνει πια. για τις επισφαλείς ε, μορφές εργασίας και η Συνομοσπονδία Συνδικάτων θα προχωρήσει και σε νέες προσπάθειες. Πρόεδρε, τελειώνω. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν με ένα συνάδελφό σας, τον Ντανιέλ Κονμπεντίτ, και υπερασπιζόμασταν το ευρώ στη Γαλλία και είχε πει το εξή ω εικόνα. Φανταστείτε ότι όλοι οι νέοι πτυχιούχοι που θα έχουν περάσει από τον έρασμο στην Τσεχία, στη Ρώμη, στο Παρίσι σε λίγα χρόνια θα πληρώσουν αφού θα έχουν ε, ε ολοκληρώσει τις σπουδέ τους επιτυχώς θα πληρώνουν το ίδιο παγωτό παντού στην Ευρώπη με το ίδιο νόμισμα, ε, ε, το ευρώ. Λοιπόν, ε, ε, αυτό χρειάζεται να δώσουμε στους νέους, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Ναι στις θυσίες, αλλά να βλέπουμε και λίγο ε, φως στην άκρη του τούνελ. Και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω, πιστεύω, πηγαίνουν ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε. Ο τελευταίος προσκεκλημένος, ειδικό είναι ο κύριος Μαξίν Τσερούτη, Διευθυντής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων στην ε, Business Europe. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξέτοιμοι βουλευτές, ε, θα μιλήσω και εγώ στα αγγλικά. Θα ήθελα αρχίζοντας να σας πω ότι η Business Europe έχει βαθιά επίγνωση της δυσχερέστατης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι και ε, είμαστε αφοσιωμένοι στην προσπάθεια εξέβρεση λύσεων, κυρίω για τη βελτίωση τη πρόσβαση των ανθρώπων στην αγορά εργασία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα υπενθυμίσω ότι το θέμα των δεξιοτήτων ε, αναδεικνύεται σταδιακά σε μία από τις βασικότερες ε, προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρούμε αυξημένο ανταγωνισμό για δεξιότητες σε ολόκληρη την παγκόσμια σκηνή. Ταυτόχρονα ε, παρατηρείται ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη ε, κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού που σχετίζεται με λόγους όπως ε, οι δημογραφικές εξελίξεις αλλά και με τα εκπαιδευτικά συστήματα ενδεχομένως δεν είναι ούτως διαμορφωμένα ώστε να αναδεικνύουν σε προτεραιότητα να καταρτίζουν και να παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες στους ανθρώπους ώστε να καλυφθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά εργασίας. Είναι επίπονη η κατάσταση με όλα αυτά τα εκατομμύρια ενέργων στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα να χειρεύουν 2 εκατομμύρια θέσει εργασία ε, που δεν πληρώνονται ακριβώ διότι ε, στην αγορά εργασία μα έχουμε ισχυρή έλλειψη σε υψηλέ δεξιότητε. Ε, τώρα, για την ανεργία, τα ποσοστά είναι τραγικά. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι σήμερα στην Ευρώπη ε, και είναι ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο κοινωνικού χαρακτήρα νομίζω πως έχει υπολογιστεί ετησίω ε, το κόστο αυτή τη ανεργία σε ένα δι ε, ευρώ. Συνιστά λοιπόν μεγάλη οικονομική πρόκληση για την Ευρώπη. Χάνεται μία γενιά ουσιαστικά και χάνοντα μία γενιά χάνουμε τη δυνατότητα αναπτυξιακή ανανέωση ε, και μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Δεν ε, μπορεί να συνεχιστεί έτσι λοιπόν αυτή η κατάσταση και ως εκ τούτου θέλουμε συγκεκριμένη δράση. Πρόεδρο, μας ζητήσατε ε, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Λοιπόν, ε, η οργάνωση Business Europe τους τελευταίους μήνες εργάζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Συστήσαμε μια task force όπου συσκέπτονται ειδικοί από διάφορες επιχειρήσεις και εξετάζουμε θέματα όπως οι μαθητής και το είδος δεξιότητων που χρειαζόμαστε ούτως ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν και να αντιστοιχούν σε και αγορέ εργασία. Ε, και τα πορίσματά μας τα καταγράψαμε μέσα σε μια έκθεση, πιστεύω ε, τα μέλη τη επιτροπή σας ε, πρώτη σημερινή συνεδρία έχουν ήδη λάβει αυτή την σύνοψη συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τι θα έπρεπε να κάνουν τα κράτη-μέλη καθώ και οι οργανώσει εργοδοτών και οι ίδιε επιχειρήσει. Παρατηρούμε πολύ μεγάλες διαφορές στην κατάσταση. Σε ορισμένε χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους, στην Ισπανία και στην Ελλάδα όπως ακούσαμε. Ε, είναι πάνω από το μέσο όρο σε πολλές χώρες ε, που τώρα εξετάζει ε, και παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργία στους νέους σε κάποιες χώρες που στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία συνδέεται με την λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί γίνεται αυτό, διότι έτσι αποκτούν εμπειρία και δεξιότητες οι νέοι που χρειάζονται για να βρουν ευκολότερα την πρώτη θέση στην αγορά εργασίας to um, look at how this good Βασισμένοι σε αυτή την παρατήρηση εξετάζουμε τις παρελθούσες εμπειρίες για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν ε, να τι χρησιμοποιήσουν οι χώρες ε, με εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται κυρίως στο σχολείο και δεν υπάρχει άσκηση σε επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει εμπειρία γιατί ε, σε αυτό εντοπίζονται και μεγαλύτερες δυσκολίες. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά τη μέσα και συγκεκριμένα συζητούσατε για τα διαρθρωτικά ταμεία προηγουμένως. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το πλέον ενδεδειγμένο συγκεκριμένα. Το Erasmus for All, το πρόγραμμα, παραδείγματο χάρη, ή τα ποσά που είναι διαθέσιμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει με πιο αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιηθούν, ώστε τα κράτη-μέλη όπου δεν λειτουργεί εύρυθμα ακόμη το εκπαιδευτικό του ε, σύστημα να ε, υποστηριχθούν και να ακολουθήσουν αυτήν την κατεύθυνση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τι εργασίε μα είναι το εξή. Σε πολλέ χώρε η επαγγελματική κατάρτιση ε, χωλαίνει διότι στην κοινή γνώμη υπάρχει πολύ αρνητική εικόνα και άρα δεν ελκύει του νέου ε, μια τέτοια προοπτική. Ίσως οι ίδιοι οι γονείς δεν εμπιστεύονται αυτήν την επαγγελματική σταδιοδρομία για για τους νέους ε, και τα παιδιά τους ε, πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να λήξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί συντονιστικά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να κάνει ότι πρέπει να βελτιώσει την εικόνα ε, της πρακτικής άσκησης της μαθητείας γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα πώς να βελτιώσουμε την εικόνα αυτής της μαγνηματικής οδού. Η κυρία Μοριγιά από την ε, επισφαλή γενιά Γενεργασιών Πρεκέρ ε, πέρασε ένα μήνυμα σαφέστατο, ε, κατέδειξε ποια είναι η κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι νέοι. Από πλευρά της δική μα οργάνωση, θα έλεγα ότι η Ευρώπη πάσχει από την γενικότερη εικόνα που έχει το επιχειρηματικό πνεύμα, ε, ε, πάσχει η ιδέα ε, της ανάληψης ιδίων πρωτοβουλίων για το μέλλον από τους νέους, για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων. Η λύση σίγουρα δεν είναι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε συνθήκες πλαίσιο, ώστε να αναπτυχθούν ιδιωτικέ πρωτοβουλίε και αυτό αρχίζει σε ατομικό επίπεδο. Ο καθένα δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη του για το μέλλον του και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση ανάπτυξη δεν είναι εφικτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διότι στη Γαλλία, ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παραδείγμα, ε, έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα από το μοντέλο οικονομικής ε, ανάπτυξης και άρα χρειάζεται ανάκτηση εμπιστοσύνη από πλευράς των επιχειρήσεων και από πλευράς ιδιωτών για να έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Χωρίς την ανάπτυξη αυτή δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε στα τωρινά επίπεδα τα επίπεδα διαβίωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, στην Ευρώπη τα κοινωνικά ε, συστήματα βασίζονται στην ε, αλληλεγγύη αλλά δεν ακολουθούνται από την απαιτούμενη οικονομική ανάπτυξη για να υποστηριχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, οπότε φτάνουμε στα σημαντικά πράγματα και ως συνήθως δεν έχουμε χρόνο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε προωθήσουμε το διάλογο και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τους δύο εισηγητέ για τον προϋπολογισμό για το 2012 και το 2013 και παρεμπιπτώς να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ γιατί ε, είναι απαραίτητη για μας αυτή η συνέχεια ανάμεσα στους δύο προϋπολογισμούς για να ορίσουμε ακριβώ τις προτεραιότητές μας και στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Τούρουνεν. Ε, σας παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι και να προσπαθήσετε ε, στις παρεμβάσεις σας ε, να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους νέους, λαμβάνοντας υπόψη και τα του προϋπολογισμού. Για ιστορικούς λόγους η κυρία Βαλσάνη ίσως να πάρει πρώτη το λόγο από τους εισηγητές. Παρακαλώ. Grazie Presidenti, e grazie a tutti i colleghi presenti per questa... Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είναι παρόντες σήμερα για αυτή τη σημερινή ακρόαση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, για αυτή την ακρόαση που είναι όχι μόνο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη λόγω τη πρόταση της Κομισιόν αλλά και γιατί προηγείται της πρόταση προπολογισμού που θα μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τα τέλη του Απριλίου. Την περασμένη χρονιά για τις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού του 2012, για τον οποίο είμαι συγκήτρια κάναμε εξ αρχής μια κοινή προσπάθεια. Και λέω κοινή προσπάθεια γιατί την αρχική μου πρόταση ως εισηγήτριας έγινε θετικά δεκτή τόσο στην Επιτροπή Προπολογισμού όσο και στις ε, ε, ειδικευμένε επιτροπές με τις οποίες συνάντησα σιγά σιγά. Για να... Έγινε λοιπόν η κοινή προσπάθεια για να τοποθετήσουμε στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού το θέμα της απασχόλησης. Της απασχόλησης σε η ίδια γραμμή με αυτόν τους, που είναι ένας από τους στόχους ε, τους πιο σημαντικούς της στρατηγικής για το 2020, ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους νέους, γιατί δυστυχώς σε την Ευρώπη που γερνά αφορά η ανεργία πολλές γενναίες, ακόμα και τις γυρεότερες που κάποτε ε, διαφορετικά <laughs> ζούσαν αυτό το πρόβλημα και ε, σίγουρα αφορά τους νέους ε, που δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, αλλά ε, σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Το θέμα της ανεργίας των νέων λοιπόν που από Τέλεσε βασικά το θέμα της καταπολέμησης ανεργίας, ήταν η μεγάλη προτεραιότητα για τον προπολογισμό του 2012 και προσπαθήσαμε να το μεταφράσουμε σε πρακτικά ζητήματα, σε, σε θετικές και χρήσιμες συνέπειες, δηλαδή όχι μόνο να είναι μια θεωρητική προτεραιότητα του, προ, του προπολογισμού, αλλά να μετατραπεί σε μια δημοσιονομική προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για προγράμματα που στόχο είχαν ακριβώς την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των νέων τελικά καταφέραμε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις που κράτησαν ολόκληρο το χρόνο, καταφέραμε να έχουμε σημαντική αύξηση ορισμένων πολύ στρατηγικών προγραμμάτων. Καταρχήν, ε, το lifelong learning, μια βίου κατάρτιση, που είναι το κλειδί της ανάπτυξης και της νεότητας, γιατί συμβολίζει όλα αυτά τα μέσα. Είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο πρόγραμμα που μας δίνει και το βαθμό στον οποίο ε, κινείται το βασικό πρόβλημα, δηλαδή συνδυασμός της καταπολέμησης της ανεργίας με τη διαθεσιμότητα μέσων για την κατάρτιση και την νέα, νέου κατάρτιση των ανθρώπων διαβίου. Ε, το lifelong learning αλλά και το εράσμο που θελήσαμε να αυξήσουμε γιατί εντός του εράσμου υπάρχει άλλο ένα κλειδί για τη λύση του προβλήματος ανεξαρτησίας. Είναι η κινητικότητα, η συγκεκριμένη δυνατότητα να κινηθεί κανείς σε διάφορες φάσεις εκμάθησης, εκπαίδευσης και όχι μόνο απασχόλησης. Και έπειτα γενικότερα το πρόγραμμα για την νεότητα. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ήταν θετική γιατί όχι μόνο μας επέτρεψε να βάλουμε περισσότερα κονδύλια σε αυτά τα προγράμματα αλλά ήταν και θετική γιατί ε, από την αρχή ε, έγινε θετικά αποδεκτό. Δηλαδή όλοι όσοι εργαζόμασταν στον προπολογισμό είχαμε την σαφή αίσθηση πως αυτά τα προβλήματα είναι ουσιαστικές προτεραιότητες και αυτό το δέχεται το Κοινοβούλιο παρότα απ' όλα αλλά και η Κομισιόν. Αυτή η προσπάθεια ωστόσο βρίσκεται στο πιο λεπτό σημείο γιατί ο προπολογισμό έχει κλείσει και πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει αυτές οι γραμμές και όλα αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να μετατραπούν σε δράση επιτόπου. Στις αρχές αυτής της ε, ακρόασης άκουσα τα λόγια του συναδέλφου Τζοβάν Λαβία που παρουσίαζε τις προτεραιότητες για το 2013 και διαπίστωσα ότι το πρόβλημα είναι πάντοτε το ίδιο, το πρόβλημα των πληρωμών. Για τη μεγάλη μου ανησυχία για, ως εισηγήτρια του 2012 ενός προπολογισμού δηλαδή που πρέπει πια να μετατραπεί σε πραγματικότητα και η δική του ανησυχία για τον Τζοβάν Λαβία για τον προπολογισμό του επόμενου έτους είναι να μην εξανεμιστεί η προσπάθεια που καταβάλλεται όταν καθορίζονται οι προτεραιότητες, όταν διαπραγματευόμαστε τον αριθμό των ε, δεσμεύσεων. Ε, να καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι κοινά αποδεκτό στο Κοινοβούλιο να υπερψηφιστεί με πλειοψηφίε προφανεί. Ε, ε Όλε αυτέ οι προσπάθειε λοιπόν να μην εξανεμιστούν και να μην ακυρώσουν τι προτεραιότητε ε, που έχουν ενταχθεί στον προπολογισμό χωρί να τι χρηματοδοτήσει. Αυτό συχνά δυστυχώ συμβαίνει με τα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει, αλλά συμβαίνει επίση γιατί οι αριθμοί είναι πολύ διαφορετικοί και με τι δράσει και με τα προγράμματα. Ανησυχία λοιπόν αφορά την κατάχρηση του μέσου της μετακίνησης των κονδυλίων που μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέσο αν πραγματικά ανταμοκρίνεται στην ανάγκη ευελιξίας του προπολογισμού, ευελιξίας ανάλογα με τις απαιτήσει και τις επίγουσες ανάγκες αλλά να μην μετατραπεί ε, προϋπολογισμός, να μην εκτροχιαστεί από τις πραγματικές του ε, στόχους και να μην ε, απαξιώσει τις γραμμές που έχουν ήδη ε, αποφασιστεί. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτές οι γραμμές του προϋπολογισμού, το lifelong learning και το εράσμος καθορίστηκαν ως προτεραιότητες γιατί θεωρήσαμε ότι πρόκειτο για προγράμματα όπου υπήρχαν ψηλότερε δυνατότητε απορρόφησης των κονδυλίων και ήμασταν βέβαιοι πω αυτέ οι γραμμέ θα μετατρέπονταν όντω σε συγκεκριμένε δράσει και δεν θα αφισβητηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, ε, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, οι πληρωμές. Θέλουμε λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια να υλοποιηθεί πραγματικά, να μετατραπεί σε δράση μέσα στο 2012. Λοιπόν, κύριε Λαβία, έτσι θα γίνουν όλα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω είπα στην προηγούμενη συζήτηση. Και όπω είπε και η συνάδελφο Μπαλτζάνη, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, χάρη στη μεγάλη όθηση που δίνει το Κοινοβούλιο, αποφάσισε να συμπεριλάβει τους νέους στις πολιτικές του προτεραιότητες. Σε φάση κρίσης, όταν η πόρη είναι πρέπει να αναζητήσουμε με κάθε τρόπο την ε, βέλτιστη χρήση των όσων έχουμε στη διάθεσή μας. Μαζιζόμενοι σε, σε κλειδιά, όπως η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των δαπανών, καθώς και σε προγράμματα και πολιτικές που αποδεικνύουν ότι έχουν μια πραγματική προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2011 εντατικοποιήσαμε τις επενδύσεις υπέρ των νέων, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν τα, οι νέοι μας αυτή την περίοδο και γιατί θεωρούμε πως τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στην οικονομική ανάκαμψη και πιο συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Ως εισηγητής για τον προπολογισμό του 2013 θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει αυτό το έργο, θα προωθήσει τις ευκαιρίες για απασχόληση, τα προγράμματα τα ενημερωτικά και θα επενδύσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Στην τελευταία σύνοδο τη Ολομέλου στο Στρασβούργο, όπω έλεγα και προηγουμένω, εγκρίναμε τι κατευθυντήριε γραμμέ για το 2013 τονίζοντας σε πολλές περιπτώσεις την ανάγκη να γίνει ειδική προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος ε, της ενεργείας των νέων, γιατί οι νέοι αποτελούν και θα αποτελούν το πιο πολύτιμο πόρο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο σύνολό της. Όπως επίσης επαναλήφθηκε στη συζήτηση στην Ολομέλη, τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. 7,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 24 ετών δεν εργάζονται και δεν σπουδάζουν και σε ορισμένες χώρες της Ένωσης φτάνουμε σε ποσοστά νεανικής ανεργίας πάνω από το 40%. Το Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία κάλεσε την Κομισιόν από το σχέδιο προπολογισμού που θα ε, παρουσιαστεί στις 25 Απριλίου να χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσουν του νέους ώστε να αναπτύξουν προσόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε απαιτήσει της αγοράς εργασίας, θα να εγγυηθεί τις δυνατότητες επαγγελματική εμπειρίας και να διευκολύνει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Νέη ανάπτυξη, καταπολέμηση της ανεργίας, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η στόχη που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντίδοτο στην κρίση για να ξαναμπεί σε κίνηση η ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά αν θέλουμε πιο μακρόπνοα να σκεφτούμε δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε και τη χρηματοδότηση του άμεσου μέλλοντος, δηλαδή μετά το 2013 και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά δύο στοιχεία φαίνεται να είναι σαφή από τώρα. Στην τελική έκθεση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Προκλήσεις στην Επιτροπή ΣΟΥΡ του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης των προγραμμάτων ε, εκπαίδευσης, κινητικότητας, νέων ε, και κατάρτισης, πέρα από τα μέτρα που έχουν οριστεί από την προσαρμογή της ε, αγοράς εργασίας. Δόθηκε επίσης μεγάλη πρωτοβουλία στην μεγάλη προτεραιότητα στην πρωτοβουλία Youth on the Move. Ένα πρόγραμμα εμβληματικό μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 ε, όπως και το Εράσμους είναι χαμηλού κόστους και κατά συνέπεια έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τέτοια προγράμματα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν μέσα στη στρατηγική του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι σαφές λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο η δράση στο Κοινοβούλιο θα είναι πάνω σε αυτές τις γραμμές που ήδη έχουν χαραχθεί. Μια δράση λοιπόν σε συνέχεια υπέρ της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Γιατί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μην ελκύσει την προσοχή των δημοσιονομικών αρχών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τουρουνούνε που ήταν η συγγητριά μας για την έκθεση πρωτοβουλίας θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους, τους ομιλήτες. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, εισηγήθηκε αυτή την πρωτοβουλία και ασχολείται με αυτό το θέμα. Ε, η ανεργία των νέων είναι ένα θέμα ιδιαίτερα, ε, είναι πηγή ανησυχίας όχι μόνο για την Επιτροπή μας αλλά για όλους και πραγματικά από την Ιανουάριο και μετά βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης και αυτό είναι μια σημαντική πρόοδο Τώρα χρειαζόμαστε χρόνο τους ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά στην πράξη και να βρούμε και τα χρήματα για να υλοποιηθούν. Αυτό δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμη. Ε, σε σχέση τώρα με την πρωτοβουλία για τους νέους κατά τη γνώμη μου μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Είναι σίγουρο δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα. Υπάρχει όντω εθνική ευθύνη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, διότι δεν έχει σχέση η λύση με το εύρο του προβλήματο που προσπαθούμε να λύσουμε. Οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει την πρωτοβουλία για τι ευκαιρίε για του νέου. Αυτό που αποφασίστηκε δηλαδή στο Συμβούλιο τον Ιανουάριο. Αφήστε τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργία. Πήραμε τα τελευταία τελευταία στοιχεία τον περασμένο μήνα πάλι αύξηση σημειώθηκε και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι σε απόγνωση όλο και περισσότερο οι νέοι δεν πιστεύουν ε, στην πολιτική την ίδια και είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά. Τέσσερα σχόλια θα κάνω, θα είμαι σύντομη όμως. Πρώτον, όλοι Όσοι ασχολούνται με την ανεργία των νέων εδώ μέσα πρέπει οπωσδήποτε να συζητούν ταυτόχρονα και την οικονομική πολιτική. Οι γενικέ διευθύνσει ε, τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή πρέπει σε ενδοϊπηρεσιακό επίπεδο να συζητούν με το έκφυν με οποιονδήποτε τι οικονομικέ πολιτικέ. Ε, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την προσφορά, πρέπει να μιλάμε και για τη ζήτηση. Να προσφερθούν νέε θέσει εργασία δηλαδή οι νέοι οι δυνατότητες που θα έχει η τωρινή γενιά είναι άμεση συνάρτηση της οικονομικής πολιτικής ε, που θα ακολουθηθεί. Οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε και νομίζω ότι η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να καταβάλει ε, ακόμη περισσότερες προσπάθειες ώστε οι οικονομικές πολιτικές να είναι υποφελείς για τους ανθρώπους και να δημιουργούν θέσεις απασχόληση όχι σε 5 και 10 χρόνια φέτος. Δεύτερον, ε, οι εγγυήσει για του νέου Youth Guarantee. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σχολίασε αυτό το επιμέρους σημείο τη έκθεσή μου και τη επιτροπή, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή αυτή την εγγύηση για του νέου, ε, μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο αυτό, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και μπορείτε να πιέσετε του υπουργού απασχόληση καθώ και του αρχηγού ε, κρατών και κυβερνήσεων. Πλησίασαν στο στόχο τον Ιανουάριο κάπω περισσότερο και είπαν ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι που βγαίνουν ναι, και τελειώνουν τι σπουδέ του θα μένουν άνεργοι κατά νότατο όριο κάποιου μήνε. Αυτό ήταν από τα συμπεράσματά του. Και τι θα κάνετε με όλου αυτού που είναι ήδη άνεργοι. Ε, δηλαδή, κοιτάζουν μπροστά και βλέπουν αυτού ε, που θα τελειώσουν τι σπουδέ του εφ' εξή. Αλλά θα κάνουμε με τα 5,5 εκατομμύρια νέου που είναι ήδη άνεργοι. Άρα, χρειαζόμαστε μια συμπληρωματική εκστρατεία. Όποιο θέλει λοιπόν να διεκδικήσει αυτή την εγγύηση για του νέου πρέπει να συνεργαστεί μαζί μα να ε, ενώσουμε τι δυνάμει είναι μας κατόπιν. Κάτι που δεν ήταν μέσα στην έκθεσή μου, αλλά παρόλα αυτά θέλω να αναφερθώ σε αυτό και νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί από όλου. Λοιπόν, το ισχυρότερο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι νέε οικονομικέ πολιτικέ, τα νέα καθεστώτα που εφαρμόζονται μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να προταθεί για την στρατηγική 2020 ένας ε, υποστόχος συγκεκριμένος ειδικό για τους νέους, δηλαδή κατά πόσο θα μειωθεί η ανεργία των νέων μέχρι το 2020 και από εκεί και πέρα θα ενταχθεί αυτό το σημείο ετησίως στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Το πέμπτο σημείο είναι αυτή, αυτός ο χάρτης ε, ε, για τις ε, ποιοτικές ε, πρακτικές ασκήσεις, ποιοτικές μαθητείες. Είναι κέρια σημασία σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με την οργάνωση Γενεγασιών και είναι με ένα εργατικό δυναμικό που δεν έχει δικαιώματα και χρησιμοποιείται και αποτελεί αντικείμενο σε δεδομένες της κατάστασης. Μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα αυτά τα μέτρα, αλλά οπωσδήποτε ε, χρειάζεται μια ε, κανονιστική ρύθμιση και γι' αυτό θα ζητήσω όχι μόνο έγγραφο εργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ε, επόμενο μήνα. Χρειαζόμαστε κάτι ισχυρότερο, συμπεράσματα του Συμβουλίου, ανακοίνωση, κάτι να μα πείτε μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, είναι κατεπήγον ίσως ε, σε πρώτο στάδιο ένα έγγραφο εργασίας, αλλά αμέσως μετά θα πρέπει να ακολουθηθεί από κάτι πιο συγκεκριμένο. Κλείνω τώρα λέγοντας ότι καλή είναι αυτή η πρωτοβουλία, αλλά σίγουρα δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερες πρωτοβουλίες, ε, ε, χρειάζεται υλοποίηση και χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών και όπως είπαν και οι δύο γενικοί συγητές για τον προϋπολογισμό, και θέλω να τους ρωτήσω κάτι, ε, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να απαντήσετε, mm. αλλά ε, στρέφουν προς τον κύριο Λαβία πόσο πιστεύετε, κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να αυξήσετε το κονδύλι για τους νέους στον προϋπολογισμό. Ξέρω ότι πρόκειται διαφορετικά κεφάλαια, διαφορετικά ταμεία, έκτε, διαβίου, εκμάθηση κτλ. Ε, είναι διαφορετικές πολιτικές, αλλά συνολικά ε, προτίθεστε εσείς να εισηγηθείτε αύξηση του συνολικού κονδυλίου και κατά πόσο και με τα χαρά να σας υποστηρίξω εγώ. Στρέφουμε τώρα προς την Επιτροπή, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε. Αυτές οι task forces ε, προσπαθούν να ανακατανύμουν τα κονδύλια. Ε, μ' αρέσει γιατί είναι μια ενεργός προσέγγιση για την ίδια τη λειτουργία των ταμείων. Χαίρομαι που εφαρμόζεται αυτή η αρχή, αλλά από πού ακριβώς ε, θα πάρετε αυτά τα κονδύλια, δεν υπάρχουν φρέσκα, από πού θα μεταφερθούν, από πού θα τα πάρετε. Δεύτερον, ε, θα ακολουθήσουν και συστάσεις για την πολιτική από αυτές τις ομάδες ε, προβληματισμού της Task Forces. Ε, ίσως έχετε περισσότερα στοιχεία και μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκουτιέρες Πιέτρο τώρα και η κυρία Αντζελίν Λί. Ακολουθούν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ούτε με αυτά που ακούω σήμερα στην Επιτροπή από την Κομισιόν. Από τότε που αρχίσαμε συζητούμε για την ενεργεία των νέων για πρώτη φορά, βλέπουμε πιο χειροπιαστά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά από τη μια λείπει η φιλοδοξία και από την άλλη περισσεύει στη γενική συζήτηση μια θολούρα. Έχουμε αργήσει. Από τη στιγμή που εντοπίσαμε το πρόβλημα και αρχίσαμε να συζητάμε την αργία των νέων εδώ μέχρι τις προτάσεις για τα πρώτα μέτρα, η κατάσταση των νέων σε κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δύσκολη. Και θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εντάξει για πρώτη φορά φέρνει τη συζήτηση και κάνει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθεί να διοργανώσει μια στρατηγική αλλά είναι κατόπιν εορτής όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε δύο λόγους ή σε δύο χρόνους. Μπορεί σήμερα να ζούμε μια κρίση και μια συγκυρία ιδιαίτερη που έχει δραματοποιήσει περισσότερο και αγωνιούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την ανεργία των νέων. Αλλά εδώ και δεκαετίες η, δεκαετία, η ανεργία συγγνώμη, των νέων είναι υπερδιπλάσια της ανεργίας γενικότερα. Και τώρα που η κρίση αυξάνει και ε, εντείνει το πρόβλημα της ανεργίας και των ε, μεγαλύτερων, ε, οι νέοι βυθίζονται στις επισφαλείς μορφές εργασίας και στην αβεβαιότητα και στην αγωνία. Τα προβλήματα είναι διορθωτικά. Και εγώ αγωνιώ πάρα πολύ για την ουσία του προγράμματος. Τι λέμε. Α, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αποσχολησιμότητα των νέων, να βρίσκουν δουλειά οι νέοι. Αλλά στα έγγραφα που φέρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μιλάει ούτε μια στιγμή για τις ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Συμφωνώ ότι έχουμε προβλήματα κατάρτισης, υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής, όπως είπε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάλειψη του σχολείου, προφανώς είναι μεγαλύτερη ενεργεία, γιατί οι είναι ακατάρτιστη. Αλλά συμφωνώ επίσης και ανησυχώ με το επιχείρημα που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, αλλά δεν λέμε πώς θα ενταχθούν, με ποιους μισθούς, ποιες ε, εισφορές, ε, ποιες αποζημιώσεις στην απόλυση. Αυτά δεν τα συζητάμε. Λέμε ότι θα κάνουμε ειδική προσπάθεια ε, για να ενθαρρύνουμε τους νέους να εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Ναι, αλλά όχι ό,τι να είναι και όχι αυτό που κάνουν πολλές χώρες στην Ευρώπη έτσι υποβόσκει ένα μήνυμα ότι οι νέοι ε, αν θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας ή δουλειά θα ζητάνε ή δικαιώματα ή εγγύησεις για δουλειά ή διεκδικήσεις. Δεν μπορεί να επιδοτούμε οποιαδήποτε θέση απασχόλησης με οποιοδήποτε κόστος και τίμημα. Δεν θέλουμε τέτοιες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ομάδα πυρογνωμόνων και την Task Force που πηγαίνει από χώρα σε χώρα κάνει μια πάρα πολύ αδιαφανή δουλειά. Όπως είπε και η κυρία Τούρινεν, υπάρχουν πολιτικές δράσεις, πολιτικοί όροι και προϋποθέσεις αυτές τις 7 χώρες ας πούμε, που πλήττονται ιδιαίτερα. Και ποιος είναι ο κοινός πανομαστής. Το Συμβούλιο λέει σε όλες αυτές τις χώρες ότι θα πρέπει να κάνουν βαθιά μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία μεταρρύθμιση που να δημιουργεί από μόνη της θέσης απασχόληση ή δημιουργεί ανάπτυξη. Απασχόληση δημιουργεί ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας τι σημαίνει, ποια είναι η ποιότητα εργασίας που δημιουργείται, πώς μπαίνει στην αγορά εργασίας, πώς διατηρείσαι και πώς βγαίνεις, με ποια δικαιώματα και με ποιες αποζημιώσεις. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ και θα ήθελα να μας πούν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν υπάρχουν και πολιτικές προϋποθέσεις και όροι ε, στις επαφές που έχουν με τις κυβερνήσεις. Γιατί ούτε από τις χώρες μας τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν μας λέει τι γίνεται εκεί πέρα. Το συζητάτε. Και για τις υποτροφίες. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε η εκπρόσωπος της επισφαλούς γενιάς, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό. Δεν μπορεί ένας νέος που να έχει καταρτιστεί, να έχει εκπαιδευτεί από το δημόσιο, να πηγαίνουν ε, μόνο επιδοτούμενοι σε κάποιε θέσεις απασχόλησης, με κάποιε υποτροφίε ή με κάποιε περιόδου άσκηση κάποια στάζ που δεν έχουν και κοινωνική ασφάλιση και είναι εξαιρετικά επισφαλή μορφή εργασίας. Υπάρχει η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και του εργαζομένου. Υπάρχει το θέμα της δημόσιας υγείας, των συστημάτων των δημοσίων και των ποιοτικών οι κοινωνικές εισφορές, ε, η κοινωνική ασφάλιση έχει νόημα. Δεν είναι ε, κάτι που περιπλέκει τη ζωή των εργαζομένων. Είναι ένα θέμα που αφορά το παρόν τους και το μέλλον τους. Ευχαριστώ πολύ. Τελείως. Ευχαριστώ κυρία Τζελίλη και μετά κύριο Στέρκας. Και σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί θέλω να ξαναδώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους μας και δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Grazie, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίως γιατί πραγματικά ασχολείστε και παρακολουθείτε, ολόκληρη η Επιτροπή παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα. Επίσης εκτίμησα την ταχύτητα με την οποία η Επιτροπή μας ε, υπέβαλε ε, ρώτηση στην Κομισιόν λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30 Ιουνίου για διευκρίνηση από πλευρά τη Κομισιόν για το πόσο σκόπευε να προγραμματίσει εκ νέου αυτά τα περίφημα 83 εκατομμύρια ευρώ ε, που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσει για την καταπολέμηση ε, της ανεργίας των νέων. Εκτιμούμε λοιπόν αυτήν ε, την πρόθεση για συνεργασία, για έλεγχο της ε, νομοθετικής πορείας, ε, της πορείας των αποφάσεων και κυρίως ε, για συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία για την λήψη των αποφάσεων. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να συνεργάζεται με την Κομισιόν και να παρακολουθεί τις εργασίες του Συμβουλίου και κυρίως των κρατών μελών προς, για παράδειγμα, αυτές τις, μιλώ για παράδειγμα για αυτή την task force όπου συμμετέχουν 8 χώρες που είναι αυτές όπου η ενεργία των νέων είναι η πιο ψηλή. Αλλά είναι ενδιαφέρον να παρακολουθείτε και η δουλειά των άλλων επτά χωρών που και αυτές αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη κατάσταση. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι ενώσεις και οι πρόσωποι των επαγγελματικών επιχειρηματικών ενώσεων γιατί χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός συμμετοχής σε αυτές τις αποφάσεις και είναι σημαντικό να ακούμε τους νέους και να συμμετέχουν οι ενώσεις των νέων σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν έκανε λόγο για διαβούλευση. Δεν κατάλαβα αν έχει ολοκληρωθεί ή αν συνεχίζεται. Ευχαριστώ θα έχει την ε, δυνατότητα να σας απαντήσει η Κομισιόν, ο κ. Σέρκας και μετά ο κ. Μάν. Ευχαριστώ. Θέλω να σας χαιρετήσω όλους και να σας καλωσορίσω. Δεν μπορώ να αναφερθώ στον καθένα ξεχωριστά. Θα επικεντρωθώ στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι σε προσωπικό βέβαια, αλλά σε θεσμικό επίπεδο. Θέλω να, να του ζητήσω ε, δύο πράγματα και να εξηγήσω γιατί τα ζητώ. Πρώτον, η σοσιαλιστική ομάδα θέλει να έχει γραπτός Ποιε είναι 7-8 χώρες που επισκεφτήκατε, ποιου είδατε και τι είπαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις χώρες. Δεν μας ενδιαφέρει η έκθεση προσωρινή. Δεν θέλουμε να δούμε τι γίνεται στη μέση του δρόμου. Το Κοινοβούλιο θέλει να είναι ε, ενεργό συμμέτοχος αυτής της προσπάθειας και όχι θεατής καθ' όλη τη διάρκεια, όχι στα, μέσα, στα μισά του δρόμου να μας ενημερώσετε. Θέλουμε γραπτός ενημέρωση. Με ποιους μιλήσατε στις χώρες αυτές, τι τους είπατε. Κάτι δεν τους δώσατε κανένα έγγραφο στις χώρες αυτές, στις αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα και η ομάδα μου θέλει να το ασκήσει, να γνωρίζει ποιοι είναι οι προσανατολισμοί που δίνεται σε αυτές τις χώρες. Δεύτερη ερώτηση και έτοιμα και αυτό τεκμηριωμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθετημένη έχει την απαραίτητη και αρκετή ευελιξία να αλλάξει τις προηγούμενες θέσεις της πριν από αυτή την άσκηση ή είναι μια άσκηση που θα γίνει ό,τι και να γίνει. Τι έγινε σήμερα το πρωί. Έχουμε δύο κόσμους. Είναι ο κόσμος των νέων που είναι στο δρόμο που διαδηλώνει τον, ε, ο κόσμος των πολιτών, ο κόσμος ε, των συνδικάτων και μετά είναι ο κόσμος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζει στον κόσμο της. 7 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη ούτε σπουδάζουν ούτε δουλεύουν. Και τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι ότι έχουμε 7 εκατομμύρια ευρώ. Πώς, τι λέει εδώ? 3 εκατομμύρια για μια μελέτη και άλλα 3 εκατομμύρια για την πρόσβαση. Δηλαδή ένα ευρώ ανά 7 εκατομμύρια νέων που δεν έχουν ούτε δουλειά ούτε σπουδές κάνουν. Λοιπόν, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Πιστεύουμε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και οι λύσεις είναι τελείως ανεπαρκείς. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Διάλογος χρειάζεται με τα κρατημέλη. Και μετά το διάλογο συστάσει, είπατε. Λόγια δηλαδή. Μα είπατε για τι εγγύσει των νέων θα κάνετε καταρτική δράση. Και θα βγάλετε διδάγματα λέτε στο τέλο του έτου και ξανά σύσταση. Και 3 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα των νέων. Κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές όπως και εκατομμύρια εκατομμύριων Ευρωπαίων που τα, αυτά τα θεωρούν μόνο αερολογίες. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα και δεν λύνεται με ασπιρίνες. Δεν είναι κρυολόγημα. Πνευμονία καραμπινάτη είναι και χρειάζονται περισσότερα από λόγια του αέρα. Γιατί θα ξαναπουδιάσουμε. Εντάξει, είναι δικά τη τα χρήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσει γιατί δεν τι αφήνουν οι Βρυξέλλες τη δημόσια χρηματοδότηση γιατί θα πρέπει όλα τα προγράμματα συστηματικά να τα περικόπτουν. Τα συμβούλια να, λιγότερο, να δίνουν λιγότερες συμβουλές στα κράτη-μέλη και περισσότερη βοήθεια παρακαλώ. Ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε συνεχίζω και συμφωνώ ε, με αυτά που είπε ο Αλεχάνδρο Σέρκας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να μην είμαστε ισχυροί μόνο στην επινόηση νέων πρωτοβολιών, αλλά Youth Opportunity Initiative λέγεται αυτό, Joy, χαρά, Ε, και θέλω να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες, δεν ξέρω γραπτός μπορείτε να μας απαντήσετε. Ποιος είναι ο κοινό μας στόχος. Youth on the move, lifelong learning, τα έχουμε ξαναπεί τόσες φορές αυτά. Σε λίγο θα μας δώσετε άλλο ένα άλλο ένα όνομα. Αυτά ε, δημιουργούν σύγχυση περισσότερο παρά λύνουν προβλήματα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα και τελικά τι θα αποκομίσουμε. Σωστά είπε η κυρία Τούρινεν. Και εγώ το είπα για τη δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών. Η εγγύηση για τους νέους λοιπόν να μην είναι κάτι το ωραίο απέναντι στον ορίζοντα να το ατενίζουμε αλλά να είναι συγκεκριμένη χειροπιαστή πρωτοβουλία. Κάποιος που δεν έχει καμία εκπαίδευση μετά από τέσσερις μήνες να του λένε ορίστε εδώ θα πας να κάνεις μαθητεία. Βέβαια αν δεν έχεις προϋποθέσεις αλλά πιο συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Και δεύτερη παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σωστά είπατε, ε, ε, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας με το οποίο εργάζομαι εγώ πολύ ε, καλά σε αγαστή συνεργασία. Το θέμα δεν είναι να παίρνουν λεφτά, να τα ε, χρησιμοποιούν ώστε να πιάνουν τόπο. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά εκείνοι που εγκαταλείπουν το σχολείο. Πώς ε, τους υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη, είναι και θέμα εκπαίδευσης. Πώς μπορούμε να έχουμε κατάρτιση για να καταλαβαίνει ο νέος ότι δεν τον αποκλείουμε αλλά τον ενσωματώνουμε. Πώς θα τον κινητροδοτήσουμε, πώς θα τον ενθαρρύνουμε, πώς θα κάνουμε τις οικογένειες που είναι μακριά από την εκπαίδευση και το σχολείο να βοηθήσουν. Γιατί συνήθω οι γονεί αφήνουν τα παιδιά του στην πόρτα του σχολείου και σου λέει ανάλαβε εσύ από εδώ και πέρα. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Εάν αυτό το συγκεκριμενοποιήσουμε θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα. Μπορείτε να μας απαντήσετε γραπτός. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Euh, Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο και θα ήθελα ε, δύο λεπτά να ακούσουμε ε, τον κάθε έναν από τους προσκεκλημένους μας για τις καταληκτικές τους παρατηρήσεις. Λοιπόν, Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Τρόικα. Ε, οπότε μπορούμε και τότε να θέσουμε, να επαναλάβουμε κάποια ερωτήματα. Ως προς τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και τα θέματα πλειοψηφίας στο Συμβούλιο υπάρχει ένα διπλό σφάλμα. Πρώτον, συνεχίζουμε να μιλάμε για την ανάπτυξη σαν να μην είχε συμβεί τίποτα το είπατε κι εσείς κυρία μου, είδαμε τα ε, στατιστικά στοιχεία για την ανάδειξη των τελευταίων ετών ε, και ε, είναι όλο ένα και ασθενέστερη η ανάδειξη, όχι μόνο λόγω της Κίνας και επειδή δεν μπορούμε να μιμηθούμε το αναπτυξιακό της πρότυπο. Φυσικά μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, αλλά αν δεν έχει δεξιότητες, τι κάνουμε, διευκολύνουμε μια ευχερή πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως μετεγκαθίστανται σε άλλες χώρε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπω προβλέπει το άρθρο 9 τη συνθήκη τη Λισαβόνα και το επαναλαμβάνω αλλά χρειάζεται για να το έχουμε κατά νου. Το άρθρο 9 μας υποχρεώνει να βελτιστοποιήσουμε την χρήση των μέσων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να, ε, για να τονώσουμε την αγορά εργασίας. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Σε αυτή την συνθήκη πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε ε, ισοδυναμεί η ανάπτυξη με το σύνολο όλων των πολιτικών λιτότητα, ώστε καν αντιλαμβάνονται ποια είναι η σημασία ε, των πολιτικών στον ε, τομέα τη ε, παιδείας, γιατί δεν μπορεί να καταμετρηθεί ποσοτικά μέσα στο σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ακόμη και στην προηγούμενη περίοδο είχαμε καλά αναπτυξιακά ποσοστά. Με 2% ισχυριζόμασταν ότι δημιουργούνται νέε θέσει στην αγορά εργασία δείτε όμως ε, τις ε, αναπτυξιακές προοπτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν μας λέτε σε κανένα σημείο ότι την επόμενη δεκαετία θα έχουμε σε οποιοδήποτε κράτος 2% ανάπτυξη. Απαντήστε λοιπόν με ποιο τρόπο θα δημιουργήσουμε θέσεις για τους νέους με ανάπτυξη κατωτέρα του 2%, ακόμη και με 2%. Το είδαμε στις προηγούμενες περιόδους, απεδείχθη ότι δεν επαρκεί αυτό για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και δεύτερον, όταν εξετάζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση συνειδητοποιούμε ότι η βασική είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε την ικανότητα να καινοτομήσουμε. Όχι για να ε, φτιάξουμε κάτι που θα μοιάζει με τους μικρούς ε, Κινέζους ε, αλλά για να επιτύχουμε ουσιαστική ανταγωνιστικότητα που όλοι το λένε αλλά κανείς δεν το κάνει. Χρειαζόμαστε ρηξικέλευτη πολιτική καινοτομία. Οι νέοι, οι νέοι θα φέρουν την καινοτομία, οι, οι γέροι θα τη φέρουν, οι νέοι, συγγνώμη δηλαδή. Αλλά ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι στις συζητήσεις μας ε, φιλάρες λέμε ότι κάνουμε και πιστεύουμε πραγματικά ότι κάνουμε κάτι αλλά είναι ε, οι ιδέες και οι προτάσεις ε, που κάνετε γιατί βασίζονται σε μια εσφαλμένη βάση. 30 ε, λεπτά μόνο κύριε Λαβία γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να ακούσουμε και τους προσκεκλημένους μας. Ναι, 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει και δύο να φύγουμε έτσι αλλιώς, γιατί έχουμε μία συνάντηση με τον Ιταλό Υπουργό. Ήθελα να δώσω μια απάντηση στην συνάδελφο Τούρουνεν που ρωτούσε τι πόρους μπορούμε να έχουμε για τα ειδικά προγράμματα υπέρ της νεότητας και της απασχόλησης των νέων. Είναι σαφές ότι θα δούμε καταρχήν στις 25 Απριλίου ποια θα είναι η πρόταση που θα υποβάλει η Κομισιόν που προετοιμάζει και τον το προσχέδιο προπολογισμού και θα μας δείξει ποια μπορεί να είναι η απορρόφηση των διαφόρων γραμμών του προπολογισμού και σε σχέση με αυτή την πρόταση ε, για τις δικές μας προτεραιότητες όπως κάναμε πέρσι και πρόπερσι ξεπεράσαμε το σχέδιο προπολογισμού για πολλές γραμμές που είχαν ε, σχέση με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, δηλαδή διαβίου ε, κατάρτιση, το έρασμα το πρόγραμμα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύω πως και φέτος αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να εστιάσουμε όσο γίνεται περισσότερους πόρους και μέσω των περιθωρίων σε αυτά τα προγράμματα που θεωρούμε προτεραιότητες για τον προπολογισμό μας. Ευχαριστώ. Ήταν σχεδόν 30 δευτερόλεπτα. Θα ξαναδώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας τώρα και θα ξεκινήσω αντίστροφα με τον κύριο Τσερούτη. Και βάζω χρονόμετρο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα είμαι σύντομος. Απαντώ σε αυτά που συζητήσατε. Ε, ε, συχνά λέμε ότι οι νέοι είναι τα πρώτα θύματα της απορρίθμισης αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Σε σχέση με αυτό Πρέπει να πω ότι στην Ευρώπη είναι διαφορετική η αγορά εργασίας από χώρα σε χώρα και οι θεσμοί της. Και σε σχέση με τα όσα βάλαμε στο έγγραφο μας για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, θα πρέπει να πούμε ότι ε, όλες οι μορφές συμβάσεων κανονικά θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ε, επιχειρηματίες να προσλαμβάνουν νέους. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Και σε σχέση με όσα είπατε, η σημασία των δικαιωμάτων και να είμαστε στο σωστό δρόμο, ε, η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία, όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς φτάνουμε στις νέες αγορές. Αυτό είναι βεβαίως εκ των όνων Και για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών που αναφέρθηκε και ως στόχος και πιστεύω ότι είναι καλός και ε, αξιέπαινος, θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δεχθούμε, να ότι τα κοινωνικά συστήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επέρχονται. Και ο μόνος τρόπος να κάνουμε τα συστήματα μας αηφόρα και βιώσιμα είναι να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, όχι να προσπαθούμε να αποτρέψουμε, να προλάβουμε τις αλλαγές και να τις εμποδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα το ξαναδούμε στο μέλλον. Αυτή θα είναι η λύση, να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Ευχαριστώ. Το λέω και στους άλλους προσκεκλημένους. Καταλάβατε ότι θα ετοιμάσουμε ε, θέσεις ε, μετά από όσα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν ειδικά σημεία για να σχολιάσετε αυτά που λέει η Κομισιόν, βεβαίως θα λάβουμε υπόψη ε, τις Δεν λέω ότι θα σας αντιγράψουμε ή ότι μας δώσετε αυτούσιο θα το επαναλάβουμε. Δεν δουλεύουμε έτσι εμείς. Ο Πατρίκ Κιλτσέρτ από το Σενεκάτα. Ευχαριστώ τέσσερις ε, παρατηρήσεις. Ε, πρώτον, δεν επιμένουμε σε αυτό. Δεν πρόκειται για συνδικάτα. Είναι ένα οικονομικό φόρουμ που καταξινομεί τις χώρες ανάλογα με την ανταγωνιστικότητά τους. Ανταδό λοιπόν κατατάσσει τι χώρε και βλέπουμε ότι στι χώρε με του υψηλότερου μισθού με την ισχυρότερη συνδικαλιστική παρουσία έχουμε ε, το, ε, ε από τα σοβαρότερα προβλήματα ανεργία. Άρα δεν δημιουργούνται έτσι οι θέσει εργασία και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ε, η διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και τι ΗΠΑ είναι ότι εκείνοι έχουν ένα τρίτο πρόγραμμα ε, ανάκαμψης. σχετικά τώρα με την στρατηγική 2020 είναι σημαντικό οι νέοι να υπάρχουν παντού σε όλα σε ολόκληρη ε, την υλοποίηση της ε, στρατηγικής και εδώ θα έλεγα ότι οι κοινωνικοί εταίροι ε, σε όλες τις χώρες όπως και οι νέοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτές τις ομάδες δράσης της Task Force ε, και θα δούμε τι συστήνεται σε επίπεδο κάθε χώρα από αυτές τις ε, ομάδες. Ε, τέλος, μαζί με την ομάδα νέων της συνομοσπονδίας μας θα καταλήξουμε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες και θα σας υποβάλουμε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πορκάρο, ευχαριστώ. Ε, ήθελα να επαναλάβω και να τονίσω κάποια από τα πράγματα που ακούσαμε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Ε, πρώτον, ε, τα θέματα απασχόλησης δεν θα λυθούν αν δεν λύσουμε το συνολικότερο πρόβλημα ανάπτυξης, άρα χρειάζεται ε, συγκεκριμένη δράση και δεύτερον ε, αυτή η εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να προβλέπεται για όλους. Χρειαζόμαστε αυτή την εγγύηση και είναι πάρα πολύ καλό που η Επιτροπή σας πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενισχύει αυτό το μήνυμα τρίτον. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ακολουθεί από μια συζήτηση σχετικά με την εναρμόνιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας στα κράτη-μέλη. Έτσι μπορεί να συντονιστούν καλύτερα οι υπόλοιπες πολιτικές με την πολιτική απασχόληση. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό και το ακούσαμε και από συναδέλφους, είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία, ένα new deal ε, για τους ε, νέους στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κάτι πιο φιλόδοξο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο πακέτο των αναπρογραμματισμένων ε, κονδυλίων Εφόσον συνιστά αυτό πολιτική προτεραιότητα για την Ένωση, πρέπει να αλλάξουμε πορεία κατά 360 μοίρες, ε, να έχουμε μια νέα φρέσκια πρόταση που ακολουθεί μια νέα κατεύθυνση και βάσει της οποίας οι νέοι είναι στο κέντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Η Φλογόνς Μογιόν τώρα για την τελευταία παρουσίαση και ίσως θα θέλατε να σχολιάσετε ε, και αυτή την πρόταση για μια εγγύηση για τους νέους Youth Guarantee που σχολίασαν διάφοροι και βλέπουμε ότι ο, εκπρόσωπο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμη δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος, ας το πούμε έτσι, δεν το σχολίασε το θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το ελάχιστο εισόδημα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Ξέρω ότι είναι πολύ διαφορετική η μισθή από χώρα σε χώρα και υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν καθόλου κατώτατο μισθό. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν μια καλή αρχή. Πέρα από την ανεργία, εκείνου που εγκαταλείπουν το σχολείο, τα κοινωνικά προβλήματα κτλ. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ελάχιστο εισόδημα. Όλο και περισσότερο λοιπόν είναι συλλογική συνείδηση το τελευταίο διάστημα Όλοι βλέπουν ότι έχουμε νέες ε, μορφές ε, κινητοποίησεων διαμαρτυριών, είδαμε τους ε, αγανακτισμένους, αλλά και άλλα κινήματα που δεν εκφράζονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιοι θύλακες αντίστασης που αρχίζουν να εκφεύγουν με τρόπο εντυπωσιακό της κρατικής εξουσίας. Από όλη την Ευρώπη φαίνεται αυτό. Και θα πρέπει να δοθεί έτσι μια δημοκρατική ορμή και να διατηρηθεί. Είναι μια οριζόντια δημοκρατία, ουσιαστική, γνήσια, άμεση. Και ε, αμφισβητούν ε, θεμελίων και βάθρων το ισχύον οικονομικό σύστημα. Και φαίνεται ότι πίσω από τους πολιτικούς ε, ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να πάρουμε εδώ το λόγο. Ε, δείχνει ότι έχετε πάρα πολύ καλή βούληση και δίνετε και το λόγο στους νέους. Ε, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το χάσμα, να ε, δοθεί συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια του κόσμου που είναι στο δρόμο που αγωνίζεται και διαμαρτύρεται. Και δυστυχώς έχει και κάποια αρνητικά, αλλά ελπίζω να ενισχυθούν τα θετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Πρόεδρος, ένα μήνυμα θα ήθελα να σας δώσω. Ε, ξέρω ότι έχετε πλήρη επίγνωση. Ως γυναίκα ε, θεωρούσα πάντα ότι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστούμε τα γυναικεία δικαιώματα είναι να ασχολούνται οι γυναίκες με αυτό. Και το ίδιο και για τους νέους. Δηλαδή, ε, εσείς να αναλάβετε τα ενία και εμείς να σας βοηθήσουμε με κάθε καλή βούληση και πνεύμα συνεργασίας. Θα δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λεπτά. Αυτή είναι η ισότητα των ευκαιριών προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για όλες τις ερωτήσεις που ήταν και πολλές τηλεγραφικά και στις προτεραιότητες της κυρίας η ε, συνολική προσέγγιση, ναι έχετε δίκιο, αλλά εάν για παράδειγμα γίνεται λόγος για την κοινωνική πολιτική, ε, αυτό είναι ένα στοιχείο μόνο ε, που θα παρουσιάσουμε ε, ε, μεταξύ άλλων τον Απρίλιο, όπως σας είπα. Δεν θα πρέπει να μπούμε στη λογική της ομάδας στόχος ε, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι, τι γίνεται με τους πιο ηλικιωμένους, τι γίνεται με τις γυναίκες, τι γίνεται με την ενεργό γύρανση. Δεν πάει έτσι. Χρειάζεται συνολική προσέγγιση. Ευρύτερη, συνολικότερη όπως ε, ζητεί και ε, ο εισηγητής σας. Κάτι άλλο. Τα αποτελέσματα ε, θα εγγραφούν απολύτως στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ας πούμε, ένα από τα πιο ορατά αποτελέσματα θα είναι οι συστάσεις που θα γίνουν προς τα κράτη-μέλη, τα οποία θα έχουν εντοπιστεί ως υπολοιπόμενα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την επαναφορά τους στον χώρο εργασίας και στην απασχόληση. Για την ενημέρωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μόνιμο διάλογο ε, με τα κράτη-μέλη, ε, Διάμεση έκθεση όχι τελική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας ενημερώνουμε διαρκώς κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διαφάνειας ή οτιδήποτε τέτοιο. Το λέγω γιατί αναφέρθηκε και από άλλους ομιλούντες του πάνελ. Συστηματικά στα κράτη-μέλη ε, συναντούσαμε ε, τους κοινωνικούς εταίρους. Για τα πιο ειδικά θέματα. Γιατί έγραφο διαβούλευσης και το χάρτη ποιότητας για τα Η πρόεδρος. Μπορώ να σας καλέσω να συνεχίσετε στα αγγλικά και να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους διερμηνείς ε, που έκαναν υπέρβαση ωραρίου. Ζητώ συγγνώμη που κάναμε διάλειμμα το πρωί και ε, το συμπληρώσαμε τώρα. Ε, στα αγγλικά βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μιλήσετε 10 λεπτά.